Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ ας ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε αρκετά σημεία στην ημερήσια διάταξη, δεν μπορούμε να καθυστερούμε. Καλώς ήρθατε και να σας υπενθυμίσω ότι στις 10.30 θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Όσοι έχουν ξεχάσει τις ηλεκτρονικές τους κάρτες, παρακαλώ να φροντίσουν να τις πάρουν. Άρχεται η συνεδρίαση. Καλημέρα σας και ας ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 2 δηλαδή. Υπάρχει μία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη εξαιτίας της αναβολής της έκθεσης Λούχαν για την υλοποίηση της ε, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής ε, για τη βελτίωση της ε, ανταγωνιστικότητας. Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη μετάφραση των 105 τροπολογιών που κατατέθηκαν για την έκθεση του κυρίου Λούχαν. Γιατί έλεγε προθεσμία αργά το βράδυ της 9ης Ιουλίου. Γι' αυτό δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη μετάφραση για να ψηφίσουμε σήμερα και ο εισηγητής ο κύριος Λούχαν ζήτησε την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συνεδρίαση της 27ης και 28ης Σεπτεμβρίου. Αν δεν έχετε αντίρρηση με αυτή την αλλαγή, την αναβολή ψηφοφορίας της Λούχαν, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Επίσης μην ξεχνάτε ότι υπάρχει απευθείας αναμετάδοση στο διαδίκτυο της συνεδρίασής μας. Σημείο 3 τώρα, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της Δευτέρας και Τρίτης Ιουνίου έχετε λάβει τα πρακτικά και ο συνήθως αν μέχρι το τέλος συνεδρίασης δεν υποβάλλετε αντιρρήσεις ή εστάσεις θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχω μερικές ανακοινώσεις. Καταρχήν, δεν βλέπω την Ουγγρική αντιπροσωπεία. Πού είναι. Α, όχι, εδώ είναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους από την Ουγγρική αντιπροσωπεία, τον κύριο Τόμας Φέλετζη, τον Υπουργό Εθνικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσόμπα Γκλένη, τον ε, ιδιαίτερο γραμματέα του Υπουργού. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Δεν ξέρω αν ε, παρήσατε κυρία Ανδρέα Χάντζερος. Εκεί πίσω. Καλώς ήρθατε κυρία Χάντζερος. Η κυρία Χάντζερος είναι επικεφαλής του τμήματος του Υπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης και κύριος Στόμας Κόβετς που είναι υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίζουμε την ε, Ουγγρική Αντιπροσωπεία δεν ε, εκδηλώσετε επιθυμία να λάβετε το λόγο, αλλά αν στη διάρκεια της συζήτησης ε, αυθόρμητα σας δημιουργηθεί αυτή η επιθυμία, πολύ ευχαρίστω. Σε ό,τι φορά τη συνεδρίαση των συντονιστών που έγινε στο Στρασβούργο, να σας πω ότι οι συντονιστές αποφάσισαν τα ακόλουθα. Καταρχήν, η Επιτροπή θα υποβάλει προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις ε, βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον της Πολιτική συνοχή. και θα ζητήσουμε συζήτηση για την προφορική ερώτηση στην πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Δεύτερη απόφαση των συντονιστών σε ό,τι αφορά το σχέδιο ψηφίσματος μετά το πέρας της συζήτησης που θα καταθέσει η Επιτροπή μας και η Γραμματεία θα το μοιράσει πριν την έκτακτη συνεδρίαση τη 6 Σεπτεμβρίου. Σχέδιο ψηφίσματος. Το σχέδιο αυτό θα αντικατοπτρίζει το έγγραφο με τις θέσεις μας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και <clears throat> θα έχουμε τις α, τροπολογίες για να ψηφίσουμε στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου το ψήφισμα. Δεύτερη προφορική ερώτηση αφορά την πολιτική στέγασης προς το Συμβούλιο. Προφορική ερώτηση. Οι συντονιστές αποφάσισαν να τη σύνταξη του κειμένου για τις δύο προφορικές ερωτήσεις και σας μοιράσαμε τα κείμενα αυτά. Επίσης εξετάσαμε τις γνωμοδοτήσεις που θα εκπονήσει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η πρώτη γνωμοδότηση αφορά τον δημοσιονομικό κανονισμό για το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη γνωμοδότηση αυτή την ανέλαβε το ΕΛΚ. Αλλά πιο συγκεκριμένα, α, ο Γιάνν Όλμπριχτ. Ο Γιάνν Όλμπριχτ θα εκπονήσει αυτή τη γνωμοδότηση. Δεύτερη γνωμοδότηση, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για, τη Βαλτική, για τον Εύξηνο Πόντο. Συγγνώμη. Για τον Εύξηνο Πόντο ε, θα συντάξει τη γνωμοδότηση ο κύριος Βίκτορ Μποστινάρου από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και η τρίτη γνωμοδότηση πέραν του ΑΕΠ και αλλαγές ε, στον κόσμο. Ε, η πράσινη, ο κύριος Ζαν θα εκπονήσει τη σχετική γνωμοδότηση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις προς τα θέματα αυτά, εγκρίνονται. Ένα άλλο ζήτημα που εξετάσαμε στους συντονιστές αφορούσε τη, σύνταξη της, ε, τη συγκρότηση μάλλον της Ειδικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις δημοσιονομικές και για μετά το 2013. Τα αρχικά της ε, ειδικής αυτής επιτροπής είναι ΣΟΥΡ. Μάλιστα η πρώτη συνεδρίαση ήδη έγινε και απαρτίζεται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 98 τον αριθμό και μάλιστα από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουμε 17 μέλη. Είναι βαρισίμαντη δηλαδή παρουσία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στη σύσταση της ειδική αυτής επιτροπής που θα επιτελέσει το έργο της μέσα στο, σε ένα έτος προκειμένου να καθορίσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά και τις προκλήσεις μετά το 2013. Θα πρέπει οι συντονιστέ να εξετάσουν πώς θα συνδυάσουμε το δικό μας έργο με το έργο αυτής της Ειδική επιτροπής και πώς θα παρακολουθήσουμε αυτό το έργο της Ειδική επιτροπής. Αυτό όμως θα το εξετάσουμε με τους συντονιστές. Αυτά ως προς το σημείο 4, τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Και περνάμε στο σημείο 5. Θα ήθελα να ξανακαλωσορίσω, γιατί τον είχαμε μαζί μα και χθε, τον κύριο Ρούντι Ντεμότ, τον Υπουργό Πρόεδρο τη Περιφέρεια Βαλονία και τη Γαλλική Κοινότητα, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου για το επόμενο εξάμεινο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος κύριε Ντεμότ που ευκαιρείτε και σήμερα για να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα εργασίας της Βελικής Προεδρίας ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για θέματα που φυσικά ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Πριν σας δώσω το λόγο όμως θα ήθελα να εκφράσω και μία ελπίδα. Ευελπιστώ ότι η εκπρόσωπος της Βελικής Προεδρίας ε, θα παρίσταται τακτικά στις συνεδριάσεις μας τους επόμενους μήνες γιατί μπαίνουμε σε μία πολύ κρίσιμη και σημαντική φάση της ε, προπαρασκευαστικής διαδικασίας, μάλλον της τελευταίας φάσης της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για την περίοδο μετά το 2013. Χωρίς άλλη χρονοτριβή θα ήθελα κύριε Ντεμότη να σας δώσω το λόγο για να ακούσουμε την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Βελγικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι ε, με ιδιαίτερη χαρά οι συνεργάτες μου, οι συναδελφοί μου θα παρακολουθήσουν του σύνεγγυη συνεργασία που κάνετε εδώ στην Επιτροπή. Επομένω, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να σα παρουσιάσω το πρόγραμμα τη Βελγική Προεδρία Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα επίση να σα παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασία όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Καταρχά, να σας πω ότι η πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ε, συνοχής αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα της Βελγικής Προεδρίας. Πολύ συχνά λέγεται ότι μία Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τοποθετείται. Δεν συστρατεύεται με τη μία την άλλη πλευρά, θέτει όμως προτεραιότητες. Το μέλλον λοιπόν της πολιτικής συνοχής για μετά την περίοδο του 2013 αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα. Για ποιο λόγο. Καταρχάς πρόκειται για ένα ζήτημα προτεραιοτήτων ατζέντα. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πέμπτη έκθεση όσον αφορά τη συνοχή. Η έκθεση αυτή θα παρέχει μία λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης. Δηλαδή, σε ποια φάση βρισκόμαστε όσον αφορά τη σύγκληση των οικονομιών μας, πώς η πολιτική συνοχή θα καταφέρει να συμβάλλει και ήδη συμβάλλει στους στρατηγικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς η πολιτική αυτή διαρθρώνεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές και με τις πολιτικές των κρατών μελών. Να κάποιες λοιπόν ανοιχτές ερωτήσεις που τίθενται, τίθενται ήδη από τώρα. Η έκθεση αυτή θα περιέχει επίσης τους πρώτους προσανατολισμούς όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2013. Ποια θα είναι η παγκόσμια αρχιτεκτονική αυτής της μελλοντικής διαρθρωτικής πολιτικής ποιες θα είναι οι στρατηγικές ε, βάσεις. Πώς θα διαρθρωθεί με την στρατηγική Ευρώπη 2020. Πώς θα καταφέρουμε να λάβουμε υπόψη μας τις νέες προκλήσεις και πιο συγκεκριμένα την πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ποιες είναι οι προτεραιότητες βάσει των οποίων η πολιτική αυτή θα επικεντρωθεί. Και τέλος, πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσων όπως τα διαφορετικά ταμεία κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Πρόεδρε, μια σημαντική προπαρασκευαστική εργασία έχει γίνει για τα ζητήματα αυτά. Πρόκειται για την ενδιάμεση έκτη έκθεση, για την πολιτική συνοχή ή ακόμα και η μελέτη περιφέρει 2020 ή θα μπορούσα να φερθώ ακόμα και στην έκθεση Μπάρκα ή στην συμβολή των προηγούμενων επιτρόπων για την περιφερειακή πολιτική και βέβαια στη δικιά σας συμβολή θα μπορούσα να αφαιρθώ κυρία Πρόεδρε. Οι υπουργοί τη περιφερειακή πολιτική έχουν ήδη αναφερθεί σε ζητήματα αυτά πολύ συχνά, είτε πρόκειται για την Μαριάνσκε Λάνσνε κατά τη διάρκεια τη τσεχική προεδρία, είτε πιο πρόσφατα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στην εργασία που έγινε από του υπουργού κατά τη διάρκεια τη Ισπανική προεδρία. Επίση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε έντονα με το ζήτημα αυτό και είπε ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να συμβάλλει πολύ έντονα στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Στις 14 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια σειρά συμπερασμάτων για την στρατηγική έκθεση 2010 όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομελίας στις 14 και 15 Απριλίου, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών ενέκριναν μία έκθεση, έκθεση του Γερμανού Μισελ Σνάιντερ, όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Τέλος, και εσείς κυρίες και κύριοι βουλευτές, εδώ και πάρα πολλούς μήνες ξεκινήσατε μια έντονη συζήτηση για το ζήτημα αυτό και καταλήξετε σε πολλά ψηφίσματα, εκ των οποίων ένα μάλιστα είδε το φως την προηγούμενη εβδομάδα, το ψήφισμα αυτό που έχει να κάνει με την ε, περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με την μάχη κατά της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, κυρίως στα πλαίσια του στόχου 2 με ιδιαίτερη προσοχή επίσης θα διαβάσω το έγγραφο τοποθέτησης το οποίο θα εγκρίνεται σήμερα, έγγραφο τοποθέτησης για την πολιτική συνοχή. Είτε πρόκειται λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε πρόκειται για το Συμβούλιο, είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε πρόκειται για τις συζητήσεις που γίνονται στις περιφέρειες της ε, πόλης, βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αναλύσουν, να σκεφτούν, να επεξεργαστούν περισσότερο την πολιτική συνοχή. Με τη δημοσίευση τη πέμπτη έκθεση για την πολιτική συνοχή κατά τη διάρκεια τη Βελγική Προεδρία, θα έχουμε πραγματικά μία καταπληκτική ευκαιρία να περάσουν πραγματικά στην ουσία του ζητήματο. Δεν πρόκειται όμω μόνο για ένα θέμα χρονοδιαγράμματο, timing θα έλεγα ότι η πολιτική συνοχή είναι καταρχάς μια πολιτική, πολιτική η οποία έχει εγγραφεί πλέον στην συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως αποτελεί μια πολύ σημαντική προτεραιότητα. Επίσης η Βελγική Προεδρία θέλει να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως η πολιτική συνοχή αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο για να πετύχουμε την ισορροπία αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περίοδου της κρίσης που διανύουμε αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχή θα καταφέρει να μας βοηθήσει να βγούμε από τις καταστροφικές συνέπειες που έχουμε δει όσον αφορά την απασχόληση και τη συνοχή. Επίσης, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 κατάφερε να καταδείξει ποιες είναι οι πραγματικές διαφορετικές αδυναμίες ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των περιφερειών, των πόλεων και γενικά των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν ένα παράγοντα μόχλευσης και μπορούν επίσης να μας δώσουν τα απαραίτητα διαρθρωτικά εργαλεία τα οποία θα καταφέρουν να μας οδηγήσουν σε ένα περιβάλλον οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης καθώς επίσης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίση, πρέπει να σα πω ότι η πολιτική συνοχή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο προκειμένου να καταφέρουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στην εσωτερική αγορά. Και βέβαια κατέχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η στρατηγική αυτή πραγματικά καλεί την ανάληψη δράσης στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν ένα πολύ σημαντικό επιχειρησιακό εργαλείο το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Για την Βελγική Προεδρία είναι πάρα πολύ σημαντικό η ενάληψη δράση Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των δραστικών ταμείων να διατηρηθεί και να ενδυναμωθεί. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να παραμείνει ένα πραγματικό παράγοντα υποστήριξη για την περιφερειακή ανάπτυξη για το σύνολο τη επικράτηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συνοχή είναι μια σημαντικότατη λοιπόν θεμελιώδη πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται σαφώ να υποστηριχθεί από το πρόγραμμα τη Βελγική Προεδρία. Η Βελγική λοιπόν Προεδρία θέλει καταρχάς να συνεχίσει το έργο που έχουν κάνει οι προηγούμενες προεδρίες και θα υποστηριχθεί ιδιαίτερα από την καταπληκτική εργασία που έχει γίνει από την Ισπανική Προεδρία και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στην έγκριση κάποιων νομοθετικών προτάσεων, οι οποίε είχαν να κάνουν με την ε, απλούστευση και την γενικότερη ρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Βελική Προεδρία θα ασχοληθεί κυρίως με την αποτελεσματικότητα της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματικά ανάγκη αυτή την πολιτική οικονομικής ανάπτυξης και αν ναι, τότε πώς θα καταφέρουμε να την εφαρμόσουμε. Προτείνουμε στα κράτη-μέλη να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση έχει να κάνει με την στοχοθέτηση θεματικών προτεραιοτήτων παρέμβασης σε συνδυασμό με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε ποια είναι τα βασικά θέματα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες όσον αφορά τη διαθρατική πολιτική και ποιους στόχους θα πρέπει να πετύχουμε. Θα πρέπει επίσης να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να οργανώσουμε αυτή την θεματοποίηση των προτεραιοτήτων. Επίσης, θα συνεργαστούμε σε στενή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους δικούς στρατηγικούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό θα θέσουμε και το ζήτημα της διάρθρωσης πολιτικής συνοχής με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα. Θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν διαφορετικοί τρόποι παρέμβασης και θα δούμε επίση πώς μπορούν οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες να εφαρμόσουν στην πράξη τι κοινοτικέ πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια καλύτερη συνέπεια και ένα καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα διαφορετικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η δεύτερη κατεύθυνση, ο δεύτερος μεγάλος προσανατολισμός, έχει να κάνει με την γεωγραφική στοχοθέτηση της πολιτικής συνοχής. Εδώ πέρα θα ασχοληθούμε κυρίως με το στόχο την, της σύγκλησης. Εφόσον διατηρήσουμε την πολιτική αυτή, θα πρέπει να δούμε για, σε ποιες περιφέρειες θα πρέπει να εφαρμοστεί και με ποιους συγκεκριμένου στόχους. Επίσης θα ασχοληθούμε και με το ζήτημα της διάρθρωσης, της διασύνθεσης της ε, πολιτικής συνοχής με την πολιτική ανταγωνιστικότητα για τις περιφέρειες και θα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορεί να διαρθρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κοινοτική χρηματοοικονομική υποστήριξη προκειμένου να ωφελήσει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Επίσης θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της αρχιτεκτονικής της πολιτικής συνοχής και πώς μπορεί αυτή να εφαρμοστεί όχι μόνο στην Ήπεθρο αλλά και στους ε, αστικούς πόλους. Θα ασχοληθούμε επίση με το ζήτημα της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Ξέρω ότι είναι ζήτημα το οποίο σας απασχόλησε ακόμη και χθε. Όλα τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση κυρίω κατά τη διάρκεια τη άτυπη συνάντηση των Υπουργών Πολιτική Συνοχή που θα λάβει χώρα στι 22 και 23 Νοεμβρίου 2010 στη Λιέγη. Συνάντηση κατά την οποία προφανώ έχω προσκαλέσει και την πρόεδρό σα, κυρία Χούμπνερ. Εφόσον το επιθυμεί η ε, Επιτροπή, όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, θα έρθω πολύ ευχαρίστως για να σας κάνω ένα απολογισμό της συνάντησης αυτής. Θα πρέπει να ασχοληθούμε επίσης και με το ζήτημα της εδαφικής συνεργασίας, να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών κοινωνικών, ε, συγγνώμη, κοινοτικών πολιτικών. Το ζήτημα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το Δεκέμβριο όταν, Ευρωπα... όταν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα εγκρίνει την στρατηγική για τον Δούναβη. Τα ζητήματα αυτά θα μας απασχολήσουν επίσης και κατά τη διάρκεια μιας συνδιάσκεψης υψηλού επίπεδου που θα λάβει η χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου στο Τουρνέ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ολοκληρώνω την παρέμβασή μου λέγοντά σα ότι θα είμαι απόλυτα διαθέσιμο απέναντι στη δική σα Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διατηρήσουμε έναν στενό διάλογο ανάμεσα στα θεσμικά μα όργανα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βασίζεστε στη Βελγική Προεδρία, η οποία θα έχει ω στόχο να διευκολύνει το διάλογο αυτό, τον διοργανικό, ανάμεσα στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και να ανοίξω τη συζήτηση. Πρώτος ο μιλητής είναι ο Λάμπερτ Φανίστελ Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είχαμε χθες συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι χρήσιμο να κάνουμε αυτό που συζητήσαμε, δηλαδή να λειτουργούμε σε διάφορα επίπεδα και, και το Βέλγιο πράγματι λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Αλλά υπάρχει ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω. Χθε μιλήσατε για το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει και τη σημασία της συνοχής σαν στοιχείο της στρατηγικής 2020 της Κομισιόν. Το θέμα λοιπόν είναι η συμμετοχή των πόλεων και των περιφερειών. Από την ατζέντα της Λισαβόνας, οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει βασίζονταν στην περιφερειακή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Είχε επιβληθεί όμως υπερβολικό άχθος ε, στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Διαπιστώσαμε ότι Το 70% των επενδύσεων ε, των ε, βιομηχανιών είναι στις ε, βιομηχανίες, γι' αυτό οι περιφέρειες ήταν καλύτερα εξοπλισμένες να αντιμετωπίσουν το θέμα. Συζητήσαμε επίσης το εδαφικό σύμφωνο του 2020 ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Την ιδέα αυτή την έχουμε προτείνει νωρίτερα, την έχουμε διαβιβάσει στον ε, Ρόμπε και στον Παρόσο και οι αντιδράσεις ήταν θετικές. Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς ότι οι συνθήκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της δομές. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε τώρα ένα νέο πενταετές πρόγραμμα, στο οποίο να λέμε ότι όσον αφορά την εφαρμογή και την χρηματοδότηση, κάθε κράτος μέλος να τα κάνει αυτά σε συνεργασία με τις πόλεις και τις περιφέρειες. Να γίνεται λοιπόν εργασία έτσι σε εθνικό επίπεδο και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά με ένα ενδεχόμενο συμβόλαιο εντό εισαγωγικών ανάμεσα στις πόλεις και τις περιφέρειες για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Ένα καλό παράδειγμα που έχουμε είναι η συμφωνία με τους δημάρχους που αποτελεί την, ε, την αυαρχίδα στο, ε, στο σύστημα αυτό. Μας ενδιαφέρει πολύ η αποτελεσματικότητα της ενέργειας. Ε, απαιτούνται πολλοί πόροι και όταν μιλάμε για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μια χρήσιμη συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή. Θα ήθελα πολύ τις δικές σας αντιδράσεις για το συλλογισμό αυτό. Μήπως θα θέλατε κιόλας να είσαστε πρέσβεις ε, της ιδέας αυτής ε, στα πλαίσια των ανοιχτών ημερών που θα έχουμε. Η κυρία Χίμπνερ είπε ότι θα πρέπει να αναφέρουμε τα σημεία κλειδιά του οράματός μας για τη συνοχή μακροπρόθεσμα. Το συζητήσαμε αυτό και χθες. Θα ήθελα όμως να μάθω εάν έχετε συνείδηση του θέματος αυτού, εάν είναι κάτι το οποίο θέλετε να θέσετε στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων του Συμβουλίου. Καλέσατε την κυρία Χίπνερ στην ε, άτυπη συνάντηση κορυφής και ήθελα να ρωτήσω ε, αν έχετε σκοπό να καλέσετε και άλλους εκπροσώπους της Επιτροπής μας ε, στα άτυπα συμβούλια. Ε, αυτό έγινε και επί Ισπανικής Προεδρίας. Ε, θα, θα ακούσουμε άλλη μια ερώτηση, η κυρία Ελίσα Πετσουρέτερ. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα ότι κυρίως θα ασχοληθείτε με θέματα της περαιτέρω εξέλιξης των διαρθρωτικών ταμείων όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή. Η σημασία έχει ποια περιφέρεια, για ποιους λόγους και από ποια ομάδα στόχο ε, θα είναι επιλέξιμη. Ε, αναφέρθηκε η χρήση του ΑΕΠ ως κριτήριο. Από τότε που η Γαλλία με την έκθεση Στίγκλης ε, ε, αμφισβήτησαν ε, το κριτήριο αυτό, υπάρχει η συζήτηση σχετικά με τον συνδυασμό του ΑΕΠ με άλλα κριτήρια. Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου του 70%, έχουν όμως με μεγάλη ανεργία ε, ε, και κοινωνικά βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Τι ρόλο παίζει η όλη αυτή η συζήτηση για τη Βελγική Προεδρία. Maybe Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμη έναν βουλευτή, ο κύριος Φρανσουά Αλφόνση. Θα συμπληρώσω αυτά που είπε η Ελίζαμπεθ. Η ομάδα μας θα ήθελε να μην είναι μοναδικό το κριτήριο του ΑΕΠ για την αξιολόγηση των πολιτικών μας, να συνοδεύεται και από άλλα. Ιδιαίτερα για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές που θα πρέπει να, να αποτελέσει προτεραιότητα της μελλοντικής μας πολιτικής, να λάβουμε υπόψη και το κριτήριο του διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε το κριτήριο όχι μόνο ΑΕΠ α, α, κατά κεφάλι της περιφέρειας, αλλά και το, τους τόνους διοξιδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν. Για παράδειγμα, εγώ κατάγομαι από νησί. Εκεί η κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακα ανά κάτοικο είναι πολύ μεγάλη εξαιτία της σημασία των μεταφορών. Άλλες περιοχές ε, που κυρίως χρησιμοποιούν άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας και εκεί θα έχουν υψηλό ποσοστό χρήσης διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί λοιπόν εκτός από το ΑΕΠ να μην έχουμε και άλλα κριτήρια ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε πολιτικές που θα μας φέρουν απτά αποτελέσματα και υπό το πρίσμα του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ελλειπής ο κατάλογος των κριτήριων. Μας λείπουν κριτήρια για την πολιτισμική άνθηση, για την βιοπικιλότητα κτλ. Νομίζω ότι και αυτά θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των μελλοντικών μας πολιτικών. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Υπουργό για να απαντήσει. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τον πρώτο αυτό γύρο ερωτήσεων και να αποτανθώ πρώτα στον κύριο Βανίλ Στερόη που ήταν και ο πρώτος που έλαβε το λόγο για να θέσει το ζήτημα της ενεργού συμμετοχής των πόλεων και των περιφερειών στη στρατηγική μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η στρατηγική που θα εφαρμόσουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία αν δεν κατορθώσουμε να βάλουμε κάποια ορόσημα σε ό,τι αφορά οι βασικούς κανόνες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ε, πόλεων και των περιφερειών. Γιατί όλα αυτά που λέμε θα μείνουν νεκρό γράμμα και πολύ αφηρημένα αν δεν εφαρμοστούν εμπράκτο από του ενδιαφερόμενους. Σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την μεταφορά των πόρων, γνωρίζουμε ότι η συνοχή στηρίζεται σε ένα βασικό θεμέλιο που είναι η βούληση να υλοποιηθούν και στην πράξη στρατηγικές. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την αρχή. ελήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες και μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών ίσως ε, δεν διαβρίναμε αρκετά το πεδίο εμβέλειας της συμμετοχής. Ίσως ε, θα πρέπει να εφοδιαστούμε και με περισσότερα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία. Νομίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ αυτής της βολονταριστικής προσέγγισης με μια μεγαλύτερη συμμετοχή και ανάμειξη όλων των ενδιαφερομένων και των εταίρων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο Βέλγιο θεσπίστηκε ένας μηχανισμός που προβλέπει ότι όλες οι ομόσπονδες οντότητες συμμετέχουν στην ε, παράλληλη εφαρμογή της στρατηγικής του 2020 με την βελική στρατηγική του 2020 με πολύ στενή παρακολούθηση. Το Σεπτέμβριο μάλιστα θα είμαστε έτοιμοι και θα έχουμε καθορίσει όλα τα στοιχεία για το πώς θα δράσουμε σε αυτές τις δύο στρατηγικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται εκ παραλλήλου. Βέβαια γνωρίζουμε θαυμάσια και τα προτερήματα και τις αδυναμίες του Βελγίου, αλλά αυτή η μετριοφροσύνη ακριβώς και τα επινοφροσύνη μάλλον μας κάνει πιο αποφασιστικούς ό,τι αφορά την συμμετοχή μας ε, ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών και την αποδοχή αυτών των πολιτικών. Και φαντάζομαι στο Συμβούλιο θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις τώρα. Κυρία Σρέτερ κύριος Αλφόνση. Σήμερα βασανιζόμαστε από πολλά ερωτηματικά, δεν θα έλεγα αμφιβολίες, αλλά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την ποσοτικοποίηση και, τη, και τον προσδιορισμό της μεταφοράς των κονδυλίων. Και διαρωτόμαστε κατά πόσο το ΑΕΠ είναι παρκές κριτήριο για να μας εξασφαλίσει μία παρακολούθηση που θα ικανοποιεί τους πάντες. Φυσικά θα πρέπει ίσως να διερευνήσουμε και άλλες ε, μεθοδολογίες και άλλους δείκτες και κριτήρια. Δεν θα αναφερθώ εδώ στη μακροοικονομική θεωρία. Αναφερθήκατε στον κύριο Σεν που ήταν βραβείο Νόμπελ Οικονομίας και άνοιξε την προοπτική και για νέους εναλλακτικού δείκτες και κριτήρια. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να, να διευρύνουμε αυτό το αναλυτικό φάσμα και για την αηφόρα ανάπτυξη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν θεωρώ ότι το διοξίδιο του άνθρακα είναι μόνο ένα στοιχείο αυτοτελές και ένα το κριτήριο, αλλά θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη και άλλοι δείκτες ίσως ε, θα μας βοηθήσουν για να δημιουργήσουμε μια πιο πλήρη εικόνα της κατάστασης. Και το κατόφλι των 75% του κυρωτικού μεσουόρου είναι επίσης ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει σε όλη τη φάση της ε, σταδιακής κατάργησης. Ακόμη λύσεις αφή δεν έχουμε, αλλά όταν κάποιος βρίσκεται στο 74% και περνάει τον πύχη και φτάνει στο 76%, όλα τα στοιχεία για την αξιολόγηση και το χαρακτηρισμό περιορίζονται στο κατόφλι και από τη στιγμή που κανείς κάποιος υπερβαίνει το κατόφλι το 75% όλα επανέρχονται στην τάξη. Τα λέω κάπως χονδρικά, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε και εναλλακτικά κριτήρια. υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, πέραν του ΑΕΠ. Το ποσοστό ανεργίας, για παράδειγμα. Ή άλλα κριτήρια, και δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω τώρα κάνοντας μια εκτενή περιγραφή. Πάντως, ε, συμμερίζομαι και εγώ τον ενθουσιασμό σας υπέρ μιας ε, ευρύτερης συζήτησης που θα λάβει υπόψη, θα προτείνει και διαφορετικά κριτήρια. Βέβαια, μια τέτοια συζήτηση θα είναι αρκετά χρονοβόρα. Και δεν θα ήθελα να δώσω την εντύπωση ότι αναφέρω μόνο θεωρίες για μακροοικονομικά θέματα, ενώ εδώ και εγώ είμαστε από άλλα πιο επίγοντα. Αν θέλουμε πάντως να εξασφαλίσουμε επιτυχή υλοποίηση των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, θα πρέπει οι δείκτες μας και τα κριτήριά μας να μην περιορίζονται στο ΑΕΠ, αλλά να είναι πιο ευρύς. Ευχαριστώ. Ο Βίκτορ Μποστινάρου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας, για τη δέσμευσή σας. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις προτεραιότητες της Βελικής Προεδρίας και στηριζόμαστε σε εσά για να προετοιμάσετε εκ των προτέρων το θεσμικό άτυπο και επίσημο πλαίσιο προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα για την πολιτική συνοχή στο μέλλον. Γνωρίζετε πολύ καλά πώς φτάσαμε στον τρέχοντα προπολογισμό, ποια ήταν η μάχη η οποία δόθηκε ανάμεσα στους υποστηρικτές της πολιτικής συνοχής και στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία συμμετείχαν σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις. Καταφέραμε πάντως να φτάσουμε σε μία λίστη, σε ένα προπολογισμό. Οι ερωτήσεις μου είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, πώς έχει η τρέχουσα κατάσταση στα πλαίσια του Συμβουλίου όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Δεύτερη ερώτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πώς θα καταφέρουν να συνεργαστούν από κοινού στα πλαίσια μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης προκειμένου να κερδίσουμε χρόνο προκειμένου να καταφέρουμε να καθορίσουμε την μελλοντική πολιτική συνοχής και προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια λύση η οποία θα είναι πολύ σημαντική, καθοριστική και απαραίτητη, δραματικά απαραίτητη θα έλεγα, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η Βελγική Προεδρία προκειμένου να προτιμάσει εκ των προτέρων τις συνθήκες και τους όρους για μια πραγματική συζήτηση που θα πρέπει να διεξαχθεί, μια συζήτηση που θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε χρόνο. Ο χρόνος πιέζει και είμαστε ήδη στο 2010. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Βίκτορ Τομάς. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μιλήσω συνέχεια των όσων υπόθηκαν. Υποστηρίζω τα όσα άκουσα από τον Υπουργό και συμφωνώ με μία από τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας, που είναι συγκεκριμένα ο χώρος της πολιτικής συνοχής μετά το 2013. Χαίρομαι που βλέπω ότι ε, τίθενται προτεραιότητες για την ε, πολιτική αυτή, προτεραιότητες οι οποίες θα συνδεθούν με την στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Παράλληλα θα ήθελα με την άδειά σας να κάνω κάποια ειρωνικά βέβαια σχόλια. Τα τελευταίους έξι μήνες δεν υπήρξε κανένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά όργανα τα οποία διόρισαν εμπειρογνώμονε, δημιούργησαν ομάδε εργασίας κτλ. Και ο ίδιο ο Επίτροπος Χάν ασχολείται προφανώς με το ζήτημα αυτό και προφανώς και η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλιστα δημιούργησε πρόσφατα μία ειδική επιτροπή για το ζήτημα αυτό και το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Προεδρίας, της Ισπανικής Προεδρίας και θα ασχοληθεί και με, την, με το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας. Και η Επιτροπή Ρέτζι, όπως σας είπα, ασχολείται πάρα πολύ με το ζήτημα. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το ακόλουθο. Η Βελγική Προεδρία έχει κάποια συγκεκριμένη ιδέα για το πώς θα καταφέρουμε να εναρμονίσουμε την εργασία που γίνεται από όλες αυτές τις επιτροπές, τις υποεπιτροπές και τις ομάδες εργασίας. γιατί μόνο καταφέρουμε να συντονίσουμε και να εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας θα οδηγηθούμε σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ ασαφή, τη στιγμή που έχουμε τόσους πολλούς παρεμβαίνοντες. Ξεχνάμε επίσης λίγο και τον Ευρωπαίο πολίτη, πιστεύω. Είναι σημαντικό να, να δούμε πώς ο επικεφαλής μιας τοπικής διοίκησης σε ένα πολωνικό χωριό, για παράδειγμα, θα είναι σε θέση να λάβει κάποιες αποφάσεις ακολουθώντας την κοινοτική πολιτική. Πώς θα οργανωθεί η πολιτική και η ζωή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αν έχουμε πολιτικές οι οποίες θα ανασαφεί σε κοινοτικό επίπεδο. Πιστεύω το σημαντικότατο είναι να έχουμε διαφάνεια και σαφήνεια σε κοινοτικό επίπεδο. Κύριο Στρεμόπουλο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε μια και μιλήσατε για βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, και θέλω να κάνω πιο συγκεκριμένα κάποια ερωτήματα που ήδη φάνηκαν από τη συζήτηση. Ε, επειδή υπάρχει μια κρίση που ιδιαίτερα κάποιες χώρες και περιοχές της ε, θίγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες, ποιοι πρέπει να είναι οι βασικοί προσανατολισμοί της περιφερειακής πολιτικής ιδιαίτερα για τις περιοχές εκείνες που έχουν πληγεί από την κρίση. Και ενώ τις χώρες της Βαλτικής, της Μεσογείου, την Ουγγαρία γνωρίζετε. Ε, αν δηλαδή θα βοηθηθούν στο να κάνουν αντικυκλική πολιτική ε, απέναντι στην κρίση και αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα βοηθηθούν στο να κάνουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που η βιωσιμότητα μπορεί να θεωρείται και πολυτέλεια, το βλέπω αυτό σε κάποιες χώρες και στη δικιά μου, αν λοιπόν μπορούν να βοηθούν στο να κάνουν επενδύσεις που να συνδέονται με τη βιωσιμότητα. Ευχαριστώ. Σας ακούμε κύριε Υπουργέ. Merci, euh, Madame la Présidente. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθώ στις παρεμβάσεις που μόλις έγιναν και να απαντήσω στον κύριο Ποσνερού όσον αφορά την θέση του Συμβουλίου και όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής πιο συγκεκριμένα. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα επίσημα τοποθετηθεί στο ζήτημα της πολιτικής αυτής. Δεν υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες ανακοινώσεις από το Συμβούλιο. Και αυτό γιατί θα συμβούν πρώτα κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε πρώτα την δημοσιονομική αξιολόγηση. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και τίθεται στα πρώτα στάδια της στρατηγικής. Καταρχάς πρέπει να δούμε με ποιους πόρους θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική και εφόσον έχουμε τους πόρους να δούμε στη συνέχεια για ποιους συγκεκριμένου στόχους. Λοιπόν, ποιοι είναι οι πόροι, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Θα αφιερώσουμε λοιπόν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να πείσουμε το Συμβούλιο για την χρησιμότητα της πολιτικής συνοχής. Και είμαι πεπισμένος, όπως ε, και πάρα πολλοί άλλοι παρατηρητές, ότι ε, δεν θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε μια οικονομική ανάπτυξη αν δεν περάσουμε πρώτα μέσω από από μια πολιτική συνοχής. Και η συνοχή σε καμία περίπτωση δεν αντιτίθεται στην οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, θα έλεγα ότι συμπληρώνει οποιαδήποτε πολιτική οικονομικής ανάπτυξης. Χωρίς πολιτική συνοχής είμαστε καταδικασμένοι να συναντήσουμε πολλές δυσκολίες. Πώς μπορούμε στην πράξη όμως να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Καταρχάς, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητε ε, συζητήσεις και να αναφερθώ και στα όσα είπε ο Τόμας Ντόιτς, ο οποίος ε, ηρωνικά αναφέρθηκε στα τόσα σεμινάρια, στι τόσες συζητήσεις, σε όλες αυτές τις αγαθές προθέσεις που ε, δηλώνουν τόσα πολλά διοικητικά όργανα όσον αφορά τη στρατηγική συνοχή. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεφύγουμε από τις ασάφεια των συζητήσεων αυτών και να ασχοληθούμε με τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Σίγουρα τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και αυτό το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε είναι η ασάφεια των μηχανισμών που χρησιμοποιούμε. Μηχανισμοί που δεν γίνονται κατανοητοί από τους πολίτες. Δεν αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στους εμπειρογνώμονες ή στην εμπειρογνωμοσύνη που μπορεί να έρθει από διάφορες πλευρές. Αναφέρομαι στους ανθρώπους που θα πρέπει να εφαρμόσουν την πολιτική αυτή. Κάθε φορά που αναφερόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να τη συμπεριλαμβάνουμε στη στρατηγική μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να διαρθρώσουμε καλύτερα τα πράγματα. Το στρατηγικό προφίλ λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ένα τέτοιο προφίλ το οποίο να γίνεται κατανοητό από τους πολίτες. Θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση, όχι απλώς μάλλον την εντύπωση, αλλά και τη βεβαιότητα προς αυτούς που καλούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε σε κοινοτικό επίπεδο, ότι τα μέτρα αυτά είναι όντως τα πιο αποτελεσματικά. Και αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Αν έχουμε τελικά μία κοινή στρατηγική και αν όντως πρέπει να εφαρμοστεί στρατηγική αυτή επιτόπου, αυτό θα γίνει. Θα σε έλεγα λοιπόν ότι ε, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγγυηθούμε το ότι στα πλαίσια μιας στρατηγικής θα ακολουθήσουμε ένα κοινό δρόμο και ότι θα μας θέσει όλοι να κερδίσουμε από τη στρατηγική αυτή. Η συντονισμένη προσπάθεια είναι σίγουρα το κλειδί της επιτυχίας. Όταν ο κύριος Βαν Ροπέι ανέλαβε την εντολή του, σε μία ανοιχτή επιστολή που έγραψε έλεγε ότι χρειάζεται μία πολύ σημαντική οριζόντια πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρθηκε στην πολιτική συνοχή λέγοντας ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει στο μέλλον να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει περισσότερο τις υπόλοιπες οριζόντιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της αρχής λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία αντίθεση ανάμεσα στις ε, κοινοτικέ ε, πολιτικές. Αυτό που γνωρίζουμε πάντως είναι το εξής, ότι αν θέλουμε η στρατηγική 2020 να αποφέρει καρπούς σε όλους τους τομείς, θα πρέπει όλοι όσοι συμβάλλουν στη στρατηγική αυτή να μπορούν να επωφελούνται όχι μόνο με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά να μπορούν να αποφεληθούν και από τα αποτελέσματα στρατηγικής αυτής. Και όντως ε, οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας φάνηκαν περισσότερο από το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φάνηκε από το ότι έχουμε μια λυσίδα με διάφορους αδύναμους κρίκους. Θα πρέπει ακριβώς αυτούς τους αδύναμους κρίκους να ενδυναμώσουμε. Στα πλαίσια λοιπόν της ε, περιφερειακής ε, πολιτικής θα πρέπει να καταφέρουμε να δούμε ποια είναι τα σημεία εστίασης, ποιες είναι οι σημαντικές προτεραιότητες επί των οποίων θέλουμε να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις. Και αφού γίνει πρώτα η δουλειά αυτή και αφού καταλάβουμε όλοι ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στα σημεία αυτά και ότι έχουμε συμφέρον να το κάνουμε, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να απομακρυνθούμε κάπως από τις επικρίσεις και τα αρωνικά σχόλια τα οποία ακούγονται σχετικά με τις ε, αόρισες συζητήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τους πιο συγκεκριμένους στόχους, και απαντώντας και στην ερώτηση του κυρίου Τρεμόπουλου, θα ήθελα να σας πω ότι ε, αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στην βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα όρο τον οποίο τον έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, χωρίς να πιστεύουμε σε αυτόν απαραίτητα. Έχει γίνει κατάχρηση του όρου αυτού. Στο μέλλον πάντως πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να δικαιωθούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε τα μέσα μας σε νέες πολιτικές. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τα απαραίτητα μέσα τα οποία έχουμε στις ε, περιφέρειες εκείνες οι οποίες ε, υστερούν θα πρέπει να καταφέρουμε πραγματικά να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια και να πετυχαίνουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να ε, συγκεντρώσουμε τους πόρους μας και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε προκειμένου να καταφέρουμε να εγκρίνουμε οριζόντιες πολιτικές σε όλες τις περιφέρειες, πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό πραγματικά βρίσκεται στο κέντρο της, του οράματος Βελγικής Προεδρίας. Είναι σημαντικό να έχουμε ως προτεραιότητα την βάσει αυτών των θεμελιωδών αξιών. Αξίες οι οποίες διέπουν την ε, περιφερειακή πολιτική. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη αν δεν έχουμε περιφέρειες οι οποίες θα μπορούν να αναλάβουν δράση μέσω μιας πολύ καλής περιφερειακής πολιτικής. Επίσης, όσον αφορά πάντα την οριζόντια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε πώς εφαρμόζονται επιμέρους πολιτικές και ποιες είναι αυτές οι οποίες επιφέρουν τη θέμενη αξία. Αναφέρομαι δηλαδή σε ένα σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης που θα μας επιτρέπει αυτή τη γίνουν επενδύσεις στα μέσα της πολιτικής συνοχής, οι επενδύσεις αυτές να αποφέρουν στη συνέχεια κέρδη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτή η βαθμολόγηση, αν θέλετε, αυτή η εποπτεία και αυτή η παρακολούθηση. Και νομίζω ότι μέσω της παρακολούθησης αποτελεσματικότητας θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε καλύτερες πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καρή Μαντελή. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και άλλες πολλές ευκαιρίες να ξανασυναντηθούμε. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος θα είναι ο ρόλος της Προεδρίας σας ή τι ρόλο θα δώσει η Προεδρία σας, η Βελική Προεδρία, στην διάσταση των πόλεων σε ό,τι αφορά το γενικό αρχιτεκτόνημα της πολιτικής συνοχής. Γιατί όπως ξέρετε στα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα το ΑΕΠ καλπάζει ενώ όλος παραδόξως οι κοινωνικές ανισότητες επίσης ε, διονγκώνονται. Πώς θα συμπεριληφθούν λοιπόν οι πόλεις στην πολιτική συνοχή σας, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας, η βελτίωση της, οικονο... της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων για παράδειγμα. Πριν από λίγο μιλήσατε για τη συμμετοχή. Όπως ξέρετε, περιμένουμε σε λίγες μέρες τη δημοσίευση των συμπερασμάτων της μεταξιολόγησης του Urban που ακριβώς ε, τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών φορέων. Εσείς μπορείτε να αξιολογήσετε την πρόοδο, αντίστοιχη πρόοδο και σε άλλα προγράμματα. Και τέλος μια ερώτηση για τη χρηστή διακυβέρνηση. Ποια είναι η θέση της Βελικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Πιστεύετε θα πρέπει να διατηρηθεί η μέθοδος αυτή, να τροποποιηθεί ή μήπως να καταργηθεί. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Η Έρικα Μάνερ. Ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε κύριε Υπουργέ, η Προεδρία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον της πολιτικής συνοχής και χαίρομαι ιδιαίτερος που ήρθατε για να συζητήσουμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να θετήσουμε μια διασταλτική ερμηνεία της πολιτικής συνοχής, μια ευρύτερη προοπτική και στο μέλλον αλλά και εν ώψη της στρατηγικής του 2020. Εγώ προσωπικά προβληματίζομαι λίγο με την αντιπαράθεση που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των στόχων της πολιτικής συνοχής και των στόχων της στρατηγικής του 2020, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Θα πρέπει να βρούμε μια διασύνδεση μεταξύ των στόχων της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής του 2020. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνέργεια των δύο πολιτικών και να υιοθετήσουμε το τρέχον επίπεδο του προπολογισμού. Γιατί αν υπάρξουν περικοπές στον προπολογισμό και αν θυγούν από, αυτέ, από αυτές οι περιφέρειες, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά και τη στρατηγική του 2020. Είναι πολύ σημαντικό για τους ηθήνοντες αυτής της πολιτικής να εξετάσουν δεόντως αυτό το θέμα. Αναφερθήκατε στην πρόσβαση στις υπηρεσίες. Χθες ο Επίτροπος ε, Ιωάννης Χάν ανέλησε πιο διεξοδικά αυτό το θέμα και είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, ευρυζωνικότητα και πρόσβαση στο διαδίκτυο όλων των περιφερειών, κάτι που θα βελτιώσει το δυναμικό των περιφερειών και θα αυξήσει τις ευκαιρίες. Θα πρέπει ακόμη και οι απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες. Αναφερθήκατε σε μία πληθώρα κριτηρίων, όπως και πολλοί συνάδελφοι, και είναι πολύ σημαντικό που και εσείς πιστεύετε ότι δεν αρκεί το ΑΕΠ και ότι ο κατάλογος των κριτηρίων θα πρέπει να διευρυνθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα στις αεροκατοικημένες περιοχές. Κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό για το μέλλον και ελπίζω να συζητηθεί στο Συμβούλιο και μάλιστα να σας ρωτήσω αν το έχετε ήδη εξετάσει. Το γεγονός ότι έχουμε έναν γυράσκοντα πληθυσμό θα δημιουργήσει ένα δημογραφικό πρόβλημα τα επόμενα 5-10 χρόνια. Κάτι που θα επηρεάσει τη συνολική κατάσταση και για την περιφερειακή πολιτική αλλά και για την πολιτική συνοχή. Καλό θα ήταν να θεσπιστούν κάποια κριτήρια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση του γυράσκοντος πληθυσμού και να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τις περιφέρειες που θα αντιμετωπίσουν τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί μια τέτοια δινή κατάσταση θα επηρεάσει και την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτά και ευχαριστώ να έχουμε και νέες ευκαιρίες στο μέλλον για να το συζητήσουμε. Δεν βλέπω τον Σον Κέλλη, έφυγε, ο Όντρεϊ Βλάσακ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ε, άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε. Χαίρομαι που για την Βελγική Προεδρία η, περιφερειακή πολιτική, η, η πολιτική συνοχή είναι ε, σημαντική προτεραιότητα. Ε, εάν χρησιμο... Ε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά του χρηματικού πόρου που έχουμε, θα πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε κάποιε περιφέρειε, ήδη εδώ και κάποια χρόνια, εισραίουν πόροι που δεν έχουν όμω αποτέλεσμα στο ΑΕΠ. Προβλέπεται έλεγχο της αποτελεσματικότητας της χρήσης ε, των ε, πόρων και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Ήδη οι παρούσες δημοσιονομικές προοπτικές καθιστούν δυνατή την ε, ανάθεση της ε, δαπάνης των πόρων ε, στο, στο κατώτερο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των πόλεων. Δεν έχουμε όμως καθόλου στοιχεία για το αν έχει λειτουργήσει καλά το σύστημα αυτό και αν θα ε, ήταν χρήσιμο να διαπληθεί η χρήση του. Όσον αφορά λοιπόν την ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση, δηλαδή την ε, επιθυμία μας να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους πόρους αυτούς, έχουμε, θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε σχέδια σχετικά με την ανάπτυξη των πόλεων. Και ήθελα να ρωτήσω εάν προβλέπετε αξιολόγηση των σχεδίων αυτών της ανάπτυξης των πόλεων. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει ε, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, ωστόσο αυτό το σύστημα των ε, ε, πιστώσεων δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως. Επίσης, όσον αφορά τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου ε, τομέα, μιλάμε δηλαδή για τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης με κάποιους ιδιωτικούς φορείς δεν έχουμε αξιολόγηση των, των συμπράξεων αυτών. Ε, προβλέπετε εσείς κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύρι... Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ως προς την ερώτηση που φάνηκε τουλάχιστον ε, σε τρεις παρεμβάσεις η αστική διάσταση της ανάπτυξης. Η λήψη υπόψη των πόλεων στην πολιτική συνοχής. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για συνοχή, για εδαφική συνοχή και για περιφερειακή πολιτική, αν αμελούμε την αστική διάσταση και το ρόλο των πόλεων ή το ρόλο των αστικών κέντρων σε αυτές τις πολιτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε την Ήπεθρο. Θα ήθελα να καθησυχάσω όσους φοβούνται κάτι τέτοιο. Απλώ θα πρέπει να έχουμε μια πολυπολική διάσταση ε, και ερμηνεία της πολιτικής συνοχή. Ό,τι αφορά την αστική διάσταση και την ε, συμπερίληψη των αστικών κέντρων στον προβληματισμό. Η πόλη σήμερα είναι ένα συμπίκνομα πολιτιστικό με τεράστιες προκλήσεις. Και όταν σήμερα μιλούμε για το θέμα της κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής, γνωρίζουμε ότι δυστυχώς στα μεγάλα κέντρα και στα προάστια τους υπάρχουν πραγματικά οξύτατες κοινωνικές διαφορές που οδηγούν σε πολύ σοβαρά προβλήματα που δεν μπορούν να παραγωνιστούν στην συνολική ανάλυση. Μην ξεχνάτε ότι η κοινωνική ένταξη, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού είναι βασική προτεραιότητα τη Βελγική προεδρία και μάλιστα θα έχουμε και ειδική εκδήλωση για το θέμα αυτό. Μία συνδιάσκεψη σε ό,τι αφορά το ρόλο του κοινωνικού ταμείου σε θέματα ένδυας και αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα γίνει στις 18 και 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, μια μικρή διαφήμιση για την εκδήλωση αυτή. Επίσης, κάτι άλλο. Η πόλη αλλά και τα προάστια δημιουργούν τεράστιες εδαφικές προκλήσεις, όχι μόνο σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας ή οικονομικής ανάπτυξης, αλλά εξορισμού αυτό το θέμα των αστικών κέντρων, της αστικοποίησης των προαστίων έχει και διασυνοριακή διάσταση και τα μείζωνα αστικά κέντρα ε, έχουν προβλήματα που ξεπερνούν το έδαφος τους. Και είναι λογικό ε, να προβληματίζεστε με τα θέματα αυτά. Είναι πολύ εύλογη η ανησυχία σας. Πάντως σας διαβεβαιώ και σας καθησυχάζω ότι η Βελική Προεδρία θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και θα διοργανώσει και ένα σχετικό σεμινάριο για να αναλυθούν όλες οι εμπειρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μεταξύ ε, του Βελγίου και της ε, Γαλλίας μεταξύ των πόλεων Κουρτρέ και Τουρνέ θα έχουμε την ανάλυση αντίστοιχου παραδείγματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αφιέρωση κάποιων οικονομικών πόρων στην, για την πολιτική μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μας κόστησε πολύ ακριβά σε θέματα οικονομικών επιλογών. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε τις οικονομικές μας επιλογές σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Το ανέφερα και για τη στρατηγική του 2020 και για την πολιτική συνοχής έχουμε το ίδιο μέλημα. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας εκεί που μπορούμε να έχουμε τα περισσότερα αποτελέσματα, τα πιο θεαματικά αποτελέσματα και σε εύλογο χρόνο να έχουμε αξιολογήσιμα και ποσοτικοποιήσιμα, μετρήσιμα αποτελέσματα, κάτι που θα δημιουργήσει και άμυλα και παράδειγμα προς για αντίστοιχους στόχους είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί. ό,τι αφορά το θέμα της δημοσιονομικής διαιτησίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά δεν έχει απεριόριστους πόρους. Και όλες οι χώρες, ακόμη και οι πιο γενναιόδορες που θέλουν να στηρίξουν μια ευρωπαϊκή πολιτική, ομοσπονδιακού χαρακτήρα, ε, είναι αρκετά απαιτητικά σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των κονδύλιων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι κονδύλια υπάρχουν στον προϋπολογισμό και τι δημοσιονομικές μάζες. Συνήθως αναφέρονται δύο. Μία, ένας σημαντικός τομέας είναι η πολιτική συνοχής. Σημαντικά κονδύλια υπάρχουν και για την πολιτική της γεωργίας. Και συνήθω αναφερόμαστε στις πολιτικές που είναι οι πιο δαπανηρές, γύρω στο 35% η καθεμία από τις δύο, και απορροφούν ένα σημαντικό τμήμα του προπολογισμού. Πάντως, μέλημα τη Βελγικής προεδρία είναι να μην ξεκινήσουμε οδυνηρές δημοσιονομικές διαιτησίες που θα μας οδηγήσουν σε αποσταθεροποιητικές καταστάσεις και αποτελέσματα. Και αυτό είπα και προηγουμένως στην ομιλία μου, προσπαθώντας να απαντήσω και σε ορισμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι διάφοροι στόχοι δεν είναι αντιφατικοί, δεν αλληλοποκλείονται σε ό,τι αφορά την ανάγκη χρηματοδότησής τους. Θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια συνέργεια μεταξύ των στόχων και να μην έχουμε ε, στόχους που να είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Ούτε θα πρέπει να ενισχύσουμε μια αντιπαλότητα της πολιτικής συνοχής με τη στρατηγική του 2020. Είναι συναφείς αυτές οι πολιτικές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η δημοσιονομική συζήτηση και πώς θα διαμορφωθεί ο προγραμματισμός. Θα τελειώσει η όλη ιστορία μετά το 2011. Πάντως εκεί μπορείτε να μας βοηθήσετε κι εσείς, γιατί εμείς θέλουμε μια επιθετική, δυναμική στάση και φυσικά να μην ξεχνούμε τους βασικούς στόχους της πολιτικής. Ό,τι αφορά τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε η ανάγκη εξασφάλισης της συμμετοχής των τοπικών φορέων και θέλουμε μια τέτοια ανάμιξη που θα μας δίνει την αίσθηση ότι βέβαια μια τέτοια ανάμειξη δεν είναι εύκολη, γιατί η ανάμειξη των τοπικών φορέων προϋποθέτει ε, να τους πείσουμε για το ότι είναι προς το συμφέρον τους μια τέτοια συμμετοχή. Επίσης, οι εθνικές δομές και οι περιφέρειες θα πρέπει να αφυπνίσουν τους τοπικούς φορείς για να τους δώσουν τα κίνητρα να συμμετέχουν και αυτή είναι η προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί μετά μια πιο ενεργός αναμίξή του. Στο θέμα της γύρασης του πληθυσμού, σίγουρα αυτή η δημογραφική πρόκληση είναι πολύ σημαντική και έχει και εδαφικές επιπτώσεις, γιατί βλέπουμε ότι η γύραση δεν είναι παρόμοια σε όλες τις χώρες. Μπορώ να σας δώσω παράδειγμα από το Βέλγιο. Η περιφέρεια των Βρυξελών δημογραφικά ανανεώνεται και ξανανιώνει, ενώ η Φλάνδρα α, ε, γυράσκει α, ε, με ταχύτερους ρυθμούς, από τη Βαλονία για παράδειγμα. Ακόμη και στην ίδια τη χώρα οι δημογραφικές προκλήσεις διαφέρουν και σκεφτείτε ότι το Βέλγιο είναι μια μικρή χώρα. Οπότε και η κατάσταση στις διάφορες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το δημογραφικό ζήτημα θα είναι διαφορετική. Και η πολιτική συνοχή θα πρέπει να, συλλα... να λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η γύρανση του πληθυσμού που είναι μια άλλη σημαντική πρόκληση πέραν της ε, αηφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως ε, βασική ανησυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι πολύ εύλογη αυτή η ανησυχία και θα πρέπει το, το δημογραφικό ζήτημα να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε μείγμα πολιτικών και φυσικά με την περιφερειακή του διάσταση. Αναφέρθηκε το θέμα του ελέγχου. Έχουμε τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Μόλις τώρα λάβαμε γνώση και ο αρμόδιος συνάδελφος προϋπολογισμού θα εξετάσει αυτή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως από άποψη της περιφερειακής ε, πολιτικής ε, ε, υπάρχει εκπεφρασμένη ανάγκη βελτίωσης των ελεκτικών μεθόδων και των επιθεωρήσεων. Γιατί αν θέλουμε αξιοπιστία θα πρέπει πρώτα να βελτιώσουμε τους ελέγχους μας. Έχουμε δύο ακόμη συναδέλφους και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ο Σον Κέλλη και η Σοφή Οκονή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να απαντήσω στο τηλέφωνο. Διότι στην εκλογική μου περιφέρεια σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι σε ατύχημα. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, είχα το προνόμιο πριν κάποιες εβδομάδες να βρεθώ στο Μανχάιμ να δω την χρηματοδότηση κάποιων ε, προγραμμάτων και ήταν μια σημαντική εμπειρία στα χρόνια μου εδώ. Ε, είδαμε να διευκολύνεται η κοινωνική ένταξη ε, με τη, τέτοια χρηματοδότηση. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσει η χρηματοδότηση σε περιοχές όπως το Μάνχαιμ και άλλες πόλεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη δική μου χώρα, ε, συνεχίζω να ασχολούμε με το πώς κατηγοριοποιούνται οι περιοχές. Ε, έχουμε την Ανατολή και τη Δύση που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και γι' αυτό σημαντικές ε, περιοχές ε, δεν λαμβάνουν τη χρηματοδότηση που θα πρέπει να έχουν. Για παράδειγμα το Λίμερικ, το οποίο είναι πολύ πιο πλούσιο το Τολίμερικ είναι πολύ πιο φτωχό από το Γκόλουεϊ, αλλά δεν λαμβάνει ε, χρηματοδότηση διότι αλλού βρίσκονται οι ε, βιομηχανίες. Ε, δεν θέλουμε λοιπόν τεχνητά και αυθαίρετα κριτήρια που να μην έχουν κανένα νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Οκονή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τι προτεραιότητε. της Βελικής Προεδρίας και την πολιτική συνοχή ω βασική προτεραιότητα και χαίρομαι που είπατε ότι είναι απαραίτητο στοιχείο της οικονομικής πολιτικής και επίκουρο, επικουρικό της οικονομικής πολιτικής και σε καμία περίπτωση πολέμιος της πολιτικής αυτής. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις διοικητικές διατυπώσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η πολιτική αυτή είναι από τις καλύτερες πολιτικές, γιατί στηρίζεται στην αλληλεγγύη και επιτρέπει μια γνήσια κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η πολιτική όμως αυτή δίνει σάρκα και οστά στην Ευρώπη, στις περιφέρειες. Γίνεται πιο ορατή στους πολίτες. Γιατί είδαμε το μεγάλο ποσοστό αποχής από τις ευρωεκλογέ κάτι που δείχνει πόσο ξένοι αισθάνονται οι πολίτες από τις, ευρω... από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η πολιτική συνοχή όμως ουσιαστικά δίνει αξιοπιστία στην Ευρώπη και πείθει τους πολίτες για το πόσο σημαντικά είναι θέματα κοινοτομίας, απασχόλησης, προβλήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητα. Η πολιτική συνοχή όμως μερικέ φορέ είναι περίπλοκη και πολύ επαχθή και αλλοιώνει την εικόνα της ε, Ευρώπης γιατί οι τοπικοί φορείς πολλέ φορέ έχουν αρνητική εντύπωση για την πολιτική συνοχή εξαιτία ε, της ε, επαχθούς γραφειοκρατίας και της περιπλοκότητας των διατυπώσεων. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να χαράξουμε μια κοινή προτεραιότητα για να απλουστεύσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτό ζητούμε και με μια σειρά εκθέσεων που έχουμε ήδη εγκρίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, η πολιτική συνοχή, όπω είπα, είναι από τι πιο ομορφε πολιτικέ και πιο ελκυστικέ πολιτικές της Ένωσης, αλλά κινδυνεύει. Διατρέχει ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο, το γνωρίζουμε όλοι, και μάλιστα ακούμε να γίνεται λόγο για κάποια σχέδια ή κάποιε απόπειρες διαμελισμού αυτής της πολιτικής, μέσω μιας παράλληλης πολιτικής των μεταφορών, μέσω μιας παράλληλης πολιτικής της απασχόλησης ε, και του κοινωνικού ταμείου. Εσείς πώς ε, προσεγγίζετε αυτό το θέμα και ποια είναι η αντίδρασή σας. Είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος στην άτυπη υπουργική συνάντηση στο Τολέδο για το στεγαστικό και εκεί είδαμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια γνήσια πολιτική κοινωνική στέγης. Εσείς ε, πώς βλέπετε την πολιτική κοινωνική στέγης για το επόμενο εξάμεινο, για την Βελική Προεδρία δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κονή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να απαντήσω καταρχάς στον κύριο Κέλλη για το ζήτημα των περιορισμών. Το θέσαμε το ζήτημα αυτό με τρεις διαφορετικές μορφές σήμερα, καταρχάς. Με τη μορφή των συντελεστών. Ποιοι είναι οι συντελεστές εκείνοι που επιτρέπουν να αξιολογήσουμε την ανάπτυξη. Είναι το ΑΕΠ, είναι το ΑΕΠ ένας ε, ικανοποιητικός συντελεστής. Η απάντηση προφανώς είναι ότι θα πρέπει να εμπλουτίσουμε τους μακροοικονομικούς συντελεστές που χρησιμοποιούμε και δεχομένως να πάμε και πέρα από τους μακροοικονομικούς αυτούς συντελεστές προκειμένου να αξιολογήσουμε πραγματικά την ανάπτυξη. Ένας δεύτερος περιορισμός ενδεχομένως έχει να κάνει με τον τρόπο παρέμβασης. Οι υφιστάμενοι τρόποι παρέμβασης στην πολιτική συνοχή δεν έχουν φτάσει τα ωριά τους. Ε, θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο προληπτικοί, προδραστικοί στη συμμετοχή της πολιτικής συνοχής. Και από ό,τι φαίνεται ότι η απάντηση είναι ότι θα μπορούσαμε όντως να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα παρέμβασης. Και έχουμε έναν τρίτο περιορισμό, τον εδαφικό περιορισμό. Πριν από λίγο αναφερθήκαμε στην ενσωμάτωση των αστικών πολιτικών, των πολιτικών για τα αστικά κέντρα. Θα πρέπει να έχουμε κάποιους εδαφικούς περιορισμούς οι οποίοι να είναι αυθαίρετοι ουσιαστικά να έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη οριοθέτηση περιοχών ή θα πρέπει πραγματικά η οριοθέτηση αυτή να γίνεται με βάση τα συγκεκριμένα προβλήματα δηλαδή να μας σε θέση να εστιάζουμε σε πιο προβληματικές περιοχές εκεί πέρα που υφίστανται πραγματικά τα προβλήματα. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες μπορούν να απέχουν μεταξύ τους μόνο κάποια χιλιόμετρα ή πόλεις οι οποίες μπορεί να βρίσκονται πολύ, διαφορετικ... πολύ μακριά η μία από την άλλη, αλλά θα πρέπει για κάθε μία από αυτές, παρά δηλαδή τη γεωγραφική ενδεχόμενη εγκύτητα, να βρισκονται πολυ πολυ μακρια διαφορετικοί συντελεστές, διαφορετικά κριτήρια. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της απλούστευσης. Έχω την εντύπωση, όπως το εξήγησα και πριν από λίγο, ότι ένα από τα δύναμα σημεία της πολιτικής μας είναι ότι ε, δεν είναι ιδιαίτερα φιλική για τους ε, χρήστες, για κάποιους χρήστες. Αν θέλουμε πραγματικά η πολιτική συνοχή να έχει μέλλον, θα πρέπει να δούμε με ποιους μηχανισμούς εφαρμόζεται στην πράξη και να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας πώς θα μπορούσαμε να διαρθρώσουμε καλύτερα την πολιτική αυτή σε τοπικό επίπεδο και το Συμβούλιο επίσης θα μπορούσε να συμβάλλει στη συζήτηση αυτή για το πώς θα καταφέρουμε να απλοποιήσουμε τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μέσω νέων νομοθεσιών, μέσω νέων κανονισμών και θα πρέπει να αποφύγουμε τις αντιφάσεις, δηλαδή να ζητάμε παράλληλα περισσότερο έλεγχο και περισσότερη απλούστευση συνάμα. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε την πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα της πολιτικής δεν σημαίνει ότι και η εφαρμογή της θα είναι αναγκαστικά πολύπλοκη. Ενδεχομένως να έχουμε μία πολύπλοκη πολιτική, η οποία όμως θα έχει τα απαραίτητα μέσα για να εφαρμοστεί με απλό τρόπο στην πράξη. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία μεγάλη ανάγκη που έχω εντοπίσει. Την ανάγκη να ασχοληθούμε με τον τρόπο εκείνο που οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές θα καταφέρουν να υποφεληθούν από τα μέσα τα οποία εμείς θεσπίσουμε σε κοινοτικό επίπεδο, γιατί και η απλούστευση περνάει μέσω των εργαλείων, μέσω των μέσων που χρησιμοποιούμε για την πολιτική συνοχή. Αν καταφέρουμε να θεσπίσουμε τα απαραίτητα εργαλεία, θα καταφέρουμε να δώσουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τοπικές αρχές και αυτό πραγματικά θα οδηγήσει σε επιτυχία. Θα ήθελα εκ μέρους όλων μας να σας ευχαριστήσω για την ανταλλαγή απόψεων αυτήν διότι μπορέσαμε να θίξουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων το οποίο ενδιαφέρει και τους συναδέλφους στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστούμε ε, για την ε, διάθεσή σας ε, να συμμετάσχετε στη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα επίσης εκ μέρους των συναδέλφων να πω ότι προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία με την Προεδρία και ελπίζουμε ότι θα μας τιμήσατε με την παρουσία σας και ότι θα καλέσετε ε, μέλη της Επιτροπής Ρέτζη στις ε, συναντήσεις που θα ε, ετοιμάσετε για την μελλοντική πολιτική. Νομίζω, συνάδελφοι, ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Προεδρία για την συνεργασία της και νομίζω ότι θα την εκφράσουμε με ένα θερμό χειροκρότημα. Uh, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από την Ουγγαρία. Είσαστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Συνάδελφοι, τώρα θα ψηφίσουμε. Και θα εκτιμούσα... Αν μπορούσαμε να ελέγξουμε αν λειτουργούν όλες οι κάρτες μας. Μπορούμε παρακαλώ λοιπόν να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Να ψηφίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Not everybody voted. Δεν ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας και φαίνεται να λειτουργεί το σύστημα. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Okay, so by the time you get it, okay. We will take into account your, hand then instead of... So we, move to point number... Ε, εντάξει, θα ψηφίσετε εσεί ε, ε, διανατάσσεω χειρό. χειρός. προχωράμε στο 6, που είναι προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμοβολίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στι αυτόνομες περιοχέ τη Μαδέρας και των, και Αζωρών. Τρει τροπολογίε έχουμε. Τροπολογία 1, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σαφώς ε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για το σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος, αρχή της ψηφοφορίας. Closed. Λήξη της ψηφοφορίας. 38 υπέρ, μία αποχή. Συν 39 υπέρ δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε. Στο σημείο 7 θα θυμάστε ε, η ψηφοφορία της έκθεσης του κύριου Λούχα αναβλήθηκε, οπότε προχωράμε στην έκθεση του Γεωργίου Σταυρακάκη για την ολοκληρωμένη θελάσσια πολιτική. Εδώ είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Έχουμε 34 τροπολογίες. Έχουμε κάποιες συμβιβαστικέ. Αρχίζουμε λοιπόν ψηφίζοντας την ε, συμβαστική τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται σαφώ. Πάμε στην τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προχωράμε στην συμβαστική τροπολογία 4, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ο κύριος Αγκουράκης, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να θεωρήσω ότι η τροπολογία μου είναι compatible με το κείμενο και γι' αυτό για λόγους και ουσίας και ιστορίας θα παρακαλούσα να τεθεί σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Έχει κάνει αντίρρηση? Εάν δεν έχει κάνει αντίρρηση να ψηφίσουμε την τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Δυστυχώς απορρίπτεται κυρία Αγκουράκη. Τροπολογία 9 υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, ε, δέκα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται να το ελέγξουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα. Να ελέγξουμε την 23 λοιπόν. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή. 24 καταπίπτει. Προχωράμε σε συμβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προχωράμε στη συμβαστική τροπολογία 4, όχι, συγγνώμη, πάμε στη συμβαστική τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 34 έχει αποσυρθεί. Να ψηφίσουμε λοιπόν για το σύνολο του σχεδίου έκθεσης. Θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 39 υπέρ. Μία ψήφος κατά και δύο αποχές. Προχωράμε τώρα. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στο θέμα 9 που είναι η έκθεση με θέμα το έργο της Ομάδας Εργασίας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Να σας θυμίσω ότι τον Νοέμβριο, στην αρχή Νοεμβρίου πέρσι, η Επιτροπή Ρέτζι αποφάσισε να δημιουργήσει την άτυπη ομάδα εργασίας με διπλό στόχο. Να παρακολουθήσει τη συνέχεια των εργασιών της ομάδας υψηλού επίπεδου που εργάζεται ε, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εξετάσει το μέλλον της, που επίσης εξετάζει το μέλλον της πολιτικής συνοχής και επίσης να ετοιμάσουν συστάσεις για την Επιτροπή ΡΕΤΖΙ για θέματα σημαντικά ε, που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις που θα λυθούν για την μελλοντική πολιτική συνοχή. Μέχρι τώρα είχαμε πέντε συναντήσεις, είχαμε ανταλλαγή απόψεων με ε, αξιωματούχους υψηλού επίπεδου της Κομισιόν που μας μίλησαν για τις συζητήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επίπεδου και με, την, ε, και με τις περιφέρειες για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Μετά από κάθε συνάντηση της ομάδας εργασίας, ε, μοιράσαμε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη τα πρακτικά των συναντήσεων. Θα ήθελα να σας πω ότι οι μήνες αυτή εργασίας ε, συζητήσεων ε, και διαπραγματεύσεων ε, οδήγησαν σε κάποια αποτελέσματα. Έχει ετοιμάσει έγγραφο θέση η ομάδα εργασίας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και το έγγραφο αυτό περιέχει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο θεμάτων που θεωρήσαμε ιδιαίτερα σημαντικά, τα οποία όμως επίσης αντικατοπτρίζουν τις θέσεις των πολιτικών ομάδων για την ε, πολιτική συνοχή στο μέλλον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα θέματα αυτά συμφωνήθηκαν από όλε τις πολιτικές ομάδες. Συμφωνήσαμε να μην μπούμε σε λεπτομέρειες στο στάδιο αυτό και συζητήσαμε το, θέμα, το έγγραφο αυτό στην συνάντηση των συντονιστών στις 21 Ιουνίου. Τελικά το οριστικοποιήσαμε, το εγκρίναμε με γραπτή διαδικασία. Την προηγούμενη Παρασκευή ε, διανύμαμε ένα έγγραφο σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΡΕΤΖΙ για να μπορούμε σήμερα να έχουμε την έγκριση του συνόλου της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ζητήσω από την Επιτροπή να εγκρίνει το έγγραφο αυτό. Δεν ξέρω, Λάμπερτ, ε, σήκωσε το χέρι σου. Θες να πάρεις το λόγο ή θέλεις απλά να υπερψηφίσεις ε, το έγγραφο. Ε, ναι, όχι, για να... Ε, επειδή συμφωνώ με το έγγραφο σήκωσα το χέρι μου, αλλά ίσως θα είναι χρήσιμο να έχουμε... Μας έδωσες μάλλον κάποιες λεπτομέρειες, αλλά οι περισσότεροι έρχονταν ακόμα βιαστικά στην αίθουσα, διότι δεν διότι σήμερα το πρωί σε 9 η ώρα μας ενημέρωσε σε σχετικά με ε, την ε, μέρα που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια. Μήπως μπορείς να επαναλάβει τι πληροφορίε αυτέ, γιατί είναι σημαντικέ οι πληροφορίε σχετικά με τη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια. Σήμερα το πρωί στις ανακοινώσει τη Προέδρου σα ενημέρωσα και σχετικά με τις ε, αποφάσεις ε, που ελήφθησαν από τους ε, συντονιστέ κατά τη τελευταία συνάντησή μα στο Στρασβούργο, όπου συμφωνήσαμε να υποβάλουμε προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τι βασικέ κατευθυντήριε γραμμέ τη βασική θέση της Κομισιόν ε, όσον αφορά τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Τη συζήτηση αυτή και την προφορική ερώτηση θέλαμε να, τις, ε, να τα έχουμε στο, στην πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Θέλαμε επίσης ε, σχέδιο ψηφίσματος η Γραμματεία πριν την έκτακτη συνεδρίασή μας στις 6 Σεπτεμβρίου θα διανύμει σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο θα αντικατοπτρίζει επακριβώς το έγγραφο θέσης ε, το οποίο θα εγκρίνουμε σήμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το έγγραφο θέσης αυτό ως βάση για το περιεχόμενο του ψηφίσματος που θέλουμε επίσης ε, να ψηφίσουμε κατά τη ε, θέση της, προσωπική, της προφορικής ερώτησης στην πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή, αμέσως ε, ε, μετά την ε, ψηφοφορία, θα σταλεί το έγγραφο θέσης στον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και στον Επίτροπο Χάν. Φυσικά θα τεθεί και στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είναι δημοσίως προσβάσιμο Καλό και εσάς να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο θέσης αυτό για να προωθήσετε τις θέσεις μας μέσω των δικών σας καναλιών. Μόλις το υπερψηφίσουμε θα είναι δημόσιο έγγραφο πια, ο Ε, η επίσημη θέση μας είναι ότι ε, θα εγκρίνουμε το, θέση μας, το έγγραφο αυτό διότι εργαστήκαμε πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ και για τη δική σας τη δουλειά. Με βάση τη διαδικασία αυτή Μπορεί στην αρχή του Σεπτεμβρίου να έχουμε κάποιες τροπολογίες, γιατί θα πρέπει να είναι επίσημο ψήφισμα εγκεκριμένο από την Ρέγι. Θα είναι ανοιχτό λοιπόν, εφόσον έχουμε πολιτική συνένεση, δεν χρειάζεται να, ξαναρχί... να τη συζήτηση για ένα σωρό λεπτομέρειες. Δεν είναι τελευταία ευκαιρία να πάρετε το λόγο, αλλά γνωρίζουμε τη διαδικασία. Γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αυτό τώρα. Και τι έγινε με τους φίλους μας ε, από τη Γεωργία που επίσης έχουν ε, μια πλήρη συζήτηση για το θέμα αυτό. Διστάζουμε κάπως να πούμε τι ακριβώς θέλουμε και πώς να το πούμε. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτήν τη γραμμή. Κανενός δεν περιορίζονται οι θέσεις ε, από αυτό, διότι θα ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο. Μια διευκρίνηση. Στις 6 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες με βάση το σχέδιο πρότασης που θα έχουμε από τη Γραμματεία που θα μετατρέψει το έγγραφο θέσης σε ψήφισμα. Κατόπιν θα έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε κατά τη δεύτερη ε, συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Τη δεύτερη η, δεύτερη θα, είναι, θα συμπίπτει με την προθεσμία για τις τροπολογίες. Ο κύριος Αγκουράκης ήθελε να πάρει το λόγο και μετά έχουμε άλλους δύο ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Όπως ε, γνωρίζετε είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας για το συγκεκριμένο έγγραφο. Διατηρούμε αυτές τις επιφυλάξεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας τρόπος αυτό να σημειωθεί. Κατά τα λοιπά, συμφωνώ με τη διαδικασία που προτείνεται και ε, επιφυλασσόμαστε για τροπολογίες το Σεπτέμβριο που θα γίνει η συζήτηση. Πάντως, ε, είναι νομίζω σημαντικό ε, η κοινή γνώμη να γνωρίζει, εφόσον πούμε ότι είναι ένα έγγραφο της Επιτροπής, ότι υπήρχαν και επιφυλάξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Angourakis. I just would like to... Ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι η πολιτική ομάδα του κυρίου Αγκουράκη αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ε, ομάδα εργασίας. Δεν συμμετείχε λοιπόν στην ε, διαδικασία αυτή την πολύμηνη. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν δεν προσυπογράφεται το έγγραφο. Σας καλούμε όμως να υποβάλλετε τις ε, ε, παρατηρήσεις σας τον Σεπτέμβριο. Επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, είναι έγγραφο της ομάδας εργασίας, δεν είναι της Επιτροπής μας. Εάν είναι έγγραφο της Επιτροπής θα πρέπει να συζητηθεί και να ψηφιστεί εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι πρόκειται για, επίσημα για έγγραφο της Επιτροπής μας. Κάνατε πολύ καλή δουλειά εσείς οι συντονιστές, ε, αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται με την προσυπογραφή. Θα το εγκρίνουμε, σημειώνουμε το περιεχόμενο δεν είναι έγγραφο της Επιτροπής μας, δεν είναι δημοκρατική διαδικασία αυτή. εργάζεται στην ομάδα εργασίας, λέτε ότι εντάξει το κλείσαμε όλο αυτό ε, και φτάνετε στην Επιτροπή και λέτε ότι πρέπει να το εγκρίνουμε. Μπορούμε να σημειώσουμε το περιεχόμενο, μπορούμε να το βάλουμε στον ιστότοπο, αλλά... Ε, δεν είναι έγγραφο της Επιτροπής. Εάν είναι έγγραφο της Επιτροπής θα πρέπει να ψηφίσουμε εδώ για κάθε σειρά του εγγράφου. Αλλιώς δεν θα συμφωνούσα ποτέ με τέτοια διαδικασία. Ζητώ συγγνώμη ε, για την αγένειά μου, αλλά νομίζω ότι στην πολιτική σας ομάδα δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας, διότι υπήρχαν σαφείς πληροφορίες τις οποίες είχαν συμφωνήσει κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας. Είχαμε τις εργασίες στην ομάδα εργασίας, Όλοι οι συντονιστέ των πολιτικών ομάδων που ήθελαν να συμμετάσχουν ήταν παρόντε. Μία πολιτική ομάδα δεν ήθελε να συμμετάσχει και συμφωνήθηκε μεταξύ των πολιτικών ομάδων ότι θα η ομάδα εργασία, δηλαδή όλε οι πολιτικέ ομάδε ε, συμφώνησαν ε, στα πλαίσια τη ομάδα εργασία. Έχετε δίκιο, δεν είναι επίσημο έγγραφο το οποίο θα ψηφίσουμε, είναι όμω έγγραφο το οποίο προσυπογράφει η Επιτροπή Ρέτζη και αποτελεί αντικείμενο συμφωνία όλων των πολιτικών ε, ομάδων. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, είναι έγγραφο το οποίο αντικατοπτρίζει τι θέσει των μελών της ομάδας Ρέτζι. Ε, δεν ξέρω ε, τι θεωρείτε ότι κάνανε οι συντονιστέ, ε, εάν ε, θεωρείτε ότι δεν συμφωνήθηκε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Θα σταλεί λοιπόν σαν έγγραφο το οποίο έχει προσυπογράψει η Επιτροπή. Αυτά είναι αυτά που συμφωνήθηκαν. Ε, ο κύριος Ποστινά. Ευχαριστώ πολύ κυρία ο κύριος Ποστινάρου, ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι ε, η ομάδα μας των σοσιαλιστών συμφωνεί απόλυτα με τη θέση σας να ψηφίσουμε το θέμα αυτό τον ε, Σεπτέμβριο και να ετοιμάσουμε ψήφισμα με βάση το έγγραφο αυτό, πράγμα που θα ενισχύσει πολύ τη θέση μας κατά τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα με τη θέση σας. Κάναμε τη δουλειά μας στην οριζόντια ομάδας, ομάδα εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Okay, so nobody else that would like to take the floor, I can... Um, Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, να θεωρήσω ότι η, επιτροπή, το, το, η πλειοψηφία της Επιτροπής προσυπογράφει το έγγραφο αυτό. Λάμπερτ. Ίσως θα ήταν σοφό να χρησιμοποιήσουμε τη γραπτή διαδικασία ώστε να είναι σαφές σε αυτούς που ακόμα έχουν αμφιβολίες σχετικά με το τι είναι, ότι τώρα σημειώνουμε την, ε, το περιεχόμενο του εγγράφου και ότι το Σεπτέμβριο θα ε, είναι ψήφισμα. Θα γίνει ψήφισμα. Μήπως μπορείτε να το, γράψετε, να το καταγράψετε αυτό, ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Το μόνο που θέλω είναι να μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος ε, της Επιτροπής προσέγραψε το έγγραφο αυτό το οποίο ετοίμασε η ομάδα εργασίας. Αν μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να προχωρήσουμε στο σημείο 10 της μερικής διάταξης. Ο Λάσλο είναι παρόν, ο Λάσλο Σούριαν δεν είναι παρόν. Τι θα κάνουμε λοιπόν, γνωρίζει κανείς αν πρόκειται να έρθει. δεν είναι παρόν. Επιτρέψτε μου να ε, αναβάλω το 10 μέχρι να έρθει ε, ο Λάσλο. Ε, να προχωρήσουμε στο θέμα 11 τη ημέσιας διάταξης που είναι εξέταση σχεδίου γνωμοδότηση του Αλέν Καντέκ για την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαίσιο έρευνας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφό μας τον κύριο Καντέκ. Συνάδελφοι, ας ακούσουμε την παρουσίαση του Αλέν Καντέκ θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής Το Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ανακοίνωση για την επλούστευση των προγραμμάτων πλαίσιο έρευνας, οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ήτρε αποφάσισαν να υποβάλουν μια έκθεση πρωτοβουλίας. Θεωρούσαν ότι μια τέτοια έκθεση αποτελεί μια έκθεση πολύ σημαντική από πολιτικής πλευράς και ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα επίπεδα έρευνας και καινοτομίας. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει την άποψή του. Η κυρία Καβάλο έγινε εισηγήτρια στην Επιτροπή Ήτρε και στις 30 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου στη συνέχεια. Ε, ζητήθηκε από τη δική μας Επιτροπή να υποβάλει μια γνωμοδότηση και αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω. Προφανώς μπορείτε να υποβάλλετε εσείς με τη σειρά σας τροπολογίε, προκειμένου να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότηση αυτή όλες τις απόψεις Επιτροπής μας και να καταφέρουμε να συμβάλλουμε στην συζήτηση που ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολιτική για την καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα, απασχόληση και προστασία του περιβάλλοντος. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 υποστηρίζει ιδιαίτερα τις ε, δραστηριότητες έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί διάφορα μέσα προκειμένου να προωθήσει την έρευνα και την ε, ανάπτυξη. Θα έλεγα ότι ε, το σημαντικότερο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης που δίνει περίπου 50 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2007-2013 για το ζήτημα της έρευνας και της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί σε επίπεδο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ πολλά προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο. Βλέπουμε όμως ότι πολλές φορές το σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Οι διαδικασίες είναι πολύ περίπλοκες, συνοδεύονται από, έναν έντονο, από ένα έντονο γραφειοκρατικό άχθος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε την έρευνα αυτή να τη μεταφράσουμε πολύ γρήγορα σε απτά αποτελέσματα. Η βελτίωση λοιπόν του όλου συστήματος υποβολής προτάσεων, μια εναρμόνιση του λογιστικού συστήματος ανάμεσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο, το να καταφέρουμε να δούμε σφαιρικά όλες τις θέσεις δαπανών όσον αφορά τα προγράμματα έρευνας και μια καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητες. Πιστεύω ότι όντως θα πρέπει να απλουστευθεί το σύστημα έγκρισης προγραμμάτων στα πλαίσια του 7ου πλαισίου έρευνας. Επίσης θα πρέπει να καταφέρουμε εκ των προτέρων να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να βασιστούμε λοιπόν στην εμπειρία που έχουμε από την πολιτική συνοχή. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ακολουθούν Οι η πολιτική συνοχή από την άλλη ακολουθούν πολλές φορές διαφορετικούς στόχους. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε υποχρεωτικά να συγκεράσουμε αυτά τα δύο προγράμματα. Η Επιτροπή μας πολύ συχνά έχει πει ότι πρέπει η πολιτική συνοχή να απλουστευτεί. Και βέβαια η συζήτηση για το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο στη συζήτηση αυτή, ιδίω στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο μετά το 2013. Θα πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για του δικαιούχου. Τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί έχουν πολλές φορές οδηγήσει σε έγκριση βέλτιστων πρακτικών στην διαχείριση των μέσων που έχουμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Θα μπορούσε λοιπόν να εμπνευστεί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στη διαχείρισή του από τα όσα έχουμε εμείς αντλήσει ως διδάγματα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και θα μπορούσε κατ' επέκταση να χρησιμοποιηθούν τα διδάγματα αυτά και στα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όπως είπε και ο συνάδελφος Λάμπερ Βανίστελ Ρόι, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών όσον αφορά το, ζήτημα, το ζήτημα της έρευνας και της ανάπτυξης. Πολλές φορές έχουμε διαφορετικά προγράμματα με διαφορετικούς στόχους, αλλά είναι σημαντικό να καταφέρουμε να πετύχουμε την απαραίτητη συνέργεια ανάμεσα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τα διαρθρωτικά ταμεία τα διαρθρωτικά ταμεία που πολλές φορές καλούνται να συγχρηματοδοτήσουν προγράμματα θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη ορατότητα, την απαραίτητη διαφάνεια προκειμένου να μπορούν να υποφεληθούν οι δικαιούχοι των ταμείων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε συμπληρωματικά προγράμματα πέρα από αυτά δηλαδή που προβλέπονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα υποβάλω μία τροπολογία προκειμένου να έχουμε μία εναρμόνιση του λογιστικού ελέγχου ανάμεσα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τα διαφορετικά ταμεία. Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ε, νομική ασφάλεια για τους δικαίουχους και θα καταφέρουμε να μειώσουμε επίσης το περιθώριο ασφάλματος το οποίο υπάρχει στα προγράμματα. Τα διαφορετικά ταμεία και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο βασίζονται σε κάποιους ε, κοινούς ε, κανόνες στην εταιρική σχέση και στη συγχρηματοδότηση. Είναι σημαντικό οι κανόνες αυτοί, οι αρχές αυτοί να τηρηθούν. Ξέρουμε επίσης στα πλαίσια τη Επιτροπής μα ότι η επιτυχία της περιφερειακής πολιτικής βασίζεται στην ανάληψη δράσης από όλους του φορείς φορεί, επίσης και στην οικονομική ασφάλεια. Στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης και του περιορισμού των δημοσίων δαπανών πιστεύω ότι η συγχρηματοδότηση θα πρέπει να γίνει ο βασικός κανόνας και ότι θα πρέπει όλοι να επιμεριστούμε τις προσπάθειες. Καλό λοιπόν όλους αυτούς που διαχειρίζονται το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο να εμπνευστούν από τις αρχές αυτές που έχουν οδηγήσει σε επιτυχία την περιφερειακή ανάπτυξη. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δεν είναι αρκετά αποκεντρωμένο όσον αφορά τις περιφέρειες. Οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτές οι οποίες εφαρμόζουν το πρόγραμμα και είναι αυτές ουσιαστικά που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι το περιφερειακό επίπεδο είναι το καλύτερο επίπεδο προκειμένου να τονώσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Ακριβώς επειδή οι περιφέρειες είναι αυτές που βρίσκονται κοντά στους δημόσιους οργανισμούς έρευνας, στα πανεπιστήμια, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, σε τοπικό επίπεδο μπορούν να δημιουργηθούν τα απαραίτητα κλάστερ, απαραίτητες ερευνητικές ομάδες που μπορούν να κάνουν βασική έρευνα αλλά και διάθεση στην αγορά των ε, αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής. Στα πλαίσια λοιπόν του 7ου προγράμματος, προγράμματος πλαίσιο θα πρέπει και τα στοιχεία αυτά να ληφθούν υπόψη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε τους στόχους του 7ου ε, αυτού προγράμματος πλαίσιο. Πιστεύω ότι ε, ο στόχος θα είναι να μπορούμε να επηρεάσουμε στην πράξη τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε δημόσιους πόρους σε προγράμματα τα οποία δεν θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ήδη επικεντρώνεται σε κάποια προγράμματα αριστείας, μεγάλης εμβέλειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τα προγράμματα αυτά θα έχουν θετική επιρροή σε όλη την κοινοτική επικράτεια Η προσέγγιση αυτή συμπληρώνει την πολιτική συνοχής που βασίζεται στην ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε μία στοχοθετημένη υποστήριξη στους πιο δυναμικούς πόλους, τους πόλους αριστείας που μπορούν να αναβαθμίσουν ουσιαστικά όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης μέσω της έρευνας που διεξάγουν. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να μας οδηγήσει στον στόχο της αριστείας και της ανταγωνιστικότητας. Η κυρία Καβάλιο επίση στην έκθεσή της ε, ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση. Λέει ότι ε, θα ήθελε να βασιστούμε περισσότερο στα από μάλλον ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην επιστημονική πλευρά, στην επιστημονική αξιολόγηση των προγραμμάτων και όχι τόσο πολύ στα αποτελέσματα. Θεωρεί ότι το να επικεντρωνόμαστε μόνο στα αποτελέσματα μπορεί να έχει μια αρνητική επίπτωση. Εγώ δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να αξιολογήσουμε τα προγράμματα με βάση τα αποτελέσματά τους. Δεν θα πρέπει παρόλα αυτά να δημιουργείται μία σύγχυση στους στόχους. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στοχεύει στην αριστεία, ενώ τα διορθωτικά ταμεία έχουν ως στόχο την εδαφική συνοχή. Και τα δύο αυτά βέβαια προγράμματα αλληλοσυμπληρώνονται. Μπορείτε λοιπόν και εσείς με τη σειρά σας μέσω τροπολογιών να συμβάλλετε στη γνωμοδότηση αυτή. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή Ήτρε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να εκφράζει καταρχάς την τοποθέτηση της δικής μας Επιτροπής, Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν τροπολογίες σας να επικεντρωθούν στον τομέα αυτό, στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης γιατί αν βγούμε από αυτό το πεδίο και υποβάλουμε τροπολογίες εκτός δικής μας αρμοδιότητας, νομίζω ότι θα αποδυναμώσουμε το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε. Είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση των σκιωδών εισηγητών, προκειμένου να καταφέρουμε να εργαστούμε επικοδομητικά για το ζήτημα αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έλα. Ε, ε, Άρχεται η συζήτηση ο κύριος Γκοτμάνης. Θα πρότεινα στον αξιότιμο εισηγητή δύο πράγματα. Το πρώτο θέμα που διαπιστώνει ε, η γνωμοδότηση είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής εκτέλεση. Φέτος, το 2010, στις πληρωμές, πληρώνουμε 30% λιγότερο λιγότερο 600 εκατομμύρια δηλαδή για την έρευνα. Επιπλέον το 2009 είχαμε 0,8% λιγότερα κονδύλια από το 2008. Και στον προϋπολογισμό το 2011 τα κονδύλια για την έρευνα θα είναι ακόμη λιγότερα από ό,τι το 2008. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ανάληψη υποχρεώσεων. Για την ανάληψη πληρωμών, ε, ανάληψη πληρωμών μιλάμε. Υπάρχει υποχρηματοδότηση και της έρευνας και του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου. Γιατί υπάρχουν ε, υποχρεώσεις και σε περιφερειακό επίπεδο για χρηματοδότηση έρευνας, αλλά άλλο υποχρεώσεις, άλλο οι πληρωμές. Δεν δίνονται τελικά αυτά τα κονδύλια, δεν γίνονται οι πληρωμές, γιατί δεν είναι έτοιμοι η αρμόδιοι των προγραμμάτων να εκταμιεύσουν αυτά τα χρήματα. Δεν υπάρχει φαίνεται καμία συνοχή και καμία συνάφεια μεταξύ του, της έρευνας και του Κοινωνικού Ταμείου, του Περιφερειακού Ταμείου με το 7ο Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο. Καμία συνεργασία, δεν υπάρχει καμία σχέση. Και μάλιστα δεν υπάρχουν έγγραφα ή δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες που να δείχνουν ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κονδυλίων συνοχής που δίνονται και από τα Περιφερειακό και ε, Κοινωνικό Ταμείο για να καλυφθούν οι ανάγκε ε, τη καινοτομία στα πλαίσια του 7ου Ερευνητικού Προγράμματο Πλαισίου. Φαίνεται ότι είναι τελείω ε, διαχωρισμένα σκέλη μεταξύ του και δεν δίνει το ένα σημασία στο άλλο. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα προβλήματα που επισημαίνουμε στην αγρομοδότηση και ίσως αυτά θα πρέπει να την παρελάβουμε και στην αγρομοδότησή μας προς την Ήτρε η κυρία Κάλεμπαχ. Ευχαριστώ θερμά. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή και η γνώμη της Επιτροπής Ρέγγι είναι πολύ σημαντικά εδώ, διότι ως Επιτροπή Περιφερειών πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας κλπ. Και σε πολλά σημεία αυτό σίγουρα αντιστοιχεί στη θέση της Επιτροπής Ήτρε. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα αρχής. Από τη μία έχουμε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Η έρευνα είναι το να κάνουμε από το χρήμα, από τις επενδύσεις γνώση, ε, ενώ η καινοτομία είναι από την γνώση να δημιουργούμε χρήμα. Ε, το θέμα λοιπόν είναι οι τόποι που βρίσκονται τα πανεπιστήμια. Σημαντικό για μένα είναι η πρόσβαση όπως ανέφερε και ο κύριος Εκαντέκ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή τα λιγότερα χρήματα εκεί δίνονται. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μικρά εργαστήρια που συνεχίζουν να έχουν τα περισσότερα προβλήματα με την γραφειοκρατία. Θέλουμε λοιπόν μια προσέγγιση που να προσανατολίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το να έχουμε μόνο μια τέτοια προσέγγιση είναι ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να δείξουμε περισσότερο ενδιαφέρον εδώ και ενδεχομένως να αναλάβουμε ε, περισσότερους, μεγαλύτερους κινδύνους. Στην Αυστρία, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διστάζουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά λόγω της ε, γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα, Εάν έχω παλιό υπολογιστή δεν μπορώ ε, εύκολα να υποβάλω τις αιτήσει για το πρόγραμμα αυτό, ενώ αν αγοράσω έναν ε, νέο υπολογιστή αυτό θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Αυτό σίγουρα αποτελεί πρόβλημα. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ο Μίκαλ Σρόιντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μπορούσα να ε, συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η συνάδελφος κάτι ε, Κάτεν Πάχτα προγράμματα. Ω προς τα προγράμματα έρευνας πάντα υπάρχουν ε, παράπονα από τους συμμετέχοντε ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσει Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω το ερώτημα Μήπω θα μπορούσαμε με μεγαλύτερη σαφήνεια από ό,τι εκφράζεται στην έκθεση της Ήτρε να ε, αναφέρουμε μια έκκληση για πιο σαφείς όρους όσον αφορά τα ε, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι για πολλές επιχειρήσεις ε, το γραφειοκρατικό άχθος είναι υπερβολικό και γι' αυτό δεν υποβάλλουν ε, αιτήσει. Θέλουμε λοιπόν μια ενιαία διαδικασία ή ένα ενιαίο πλαίσιο για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, άσχετα από το αν μιλάμε για πρόγραμμα πλαίσιο ε, έρευνας, ε, για ε, προγράμματα των διαφορετικών και περιφερειακών ταμείων. Κυρία Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρότασή του. Έχω κάποιες παρατηρήσεις ε, που θα τις ε, υποβάλω και ως τροπολογίες κάποια στιγμή. Καταρχήν θεωρώ ότι θα πρέπει η γνωμοδότηση αυτή να επικεντρωθεί σε μία από τις προτεραιότητές μας για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Δηλαδή στην ε, αισθητή αύξηση των κονδυλίων για την καινοτομία, ιδιαίτερα στον τομέα της αηφόρου ανάπτυξης και για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας, για τις ανανεώσιμες ενέργειες, για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτίριων. Όλα αυτά για να προετοιμάσουμε όλες, όλους τους προσανατολισμούς περί καινοτομίας και να προτρέξουμε κατά κάποιο τρόπο για να προλιάνουμε το έδαφος για μια πιο έξυπνη, για πιο αηφόρο καινοτομία με συγκεκριμένο όμως ε, πρόσωπο για να έχουμε αυτά αποτελέσματα αυτής της καινοτομίας. Να λάβουμε υπόψη όλα τα νέα δεδομένα. Την ε, περιβαλλοντική επίπτωση αλλά και την κοινωνική επίπτωση. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον κόσμο που μας ε, τριγυρίζει αν δεν αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες που πρέπει να, αντιμετωπίσουν, να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Όλες αυτές οι αναταραχές εξαιτής παγκοσμιοποίησης, το δημογραφικό πρόβλημα και όλα αυτά μας φέρουν στο επίκεντρο την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία και στις επιχειρήσεις. Προσοχή όμως, αν θέλουμε να, αντιληφθούμε τον κόσμο μας σήμερα, τον κόσμο στον οποίο ζούμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη γνώμη των ιστορικών, των κοινωνιολόγων. Και αυτοί έχουν το ρόλο τους, ας μην τους ξεχνούμε. Δυστυχώς ε, δεν βλέπω να υπάρχει στην γνωμοδότηση ο συσχετισμός μεταξύ καινοτομία και κοινωνικής ένταξης. Είναι απαραίτητο να συνδυάσουμε τη συνοχή και την ανάπτυξη με μια ολοκληρωμένη κοινωνική προσέγγιση. Κάτι που υπάρχει στα κοινοτικά προγράμματα in Europe. Και βασικό στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να υποστηρίξουν την καινοτομία στις μειονεκτούσες περιοχές ή σε στρώματα μειονεκτούντα του πληθυσμού σε, στις πόλεις και θα πρέπει το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο να συμβάλλει σε αύξηση του, της πρόσβασης στην παιδεία ή στην κατάρτιση κάποιων ευπαθών στρωμάτων του πληθυσμού ή να μας βοηθήσει να περιορίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες στις πόλεις και στις περιφέρειες να βελτιώσουμε την κινητικότητα ή την πρόσβαση στον εξοπλισμό. Πολλά μπορούν να γίνουν απτά πράγματα από το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο και θα σας τα υποβάλω και με τη μορφή τροπολογιών. Και μακάρι να τις λάβετε υπόψη, γιατί πιστεύω ότι σήμερα η έρευνα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο και να ακούσουμε και τους ερευνητές μας, το ΣΕΝΕΡΕΣ, το γνωρίζετε, όπως και εγώ, ή τώρα ή ποτέ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντέλη. Δεν ξέρω... Α, ο Σον ο Πολύ σύντομα. Καταρχήν να επενέσω τον Αλέν για την έκθεσή του. Κάποιες παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι η η ιδέα του να βασίζεται η καινοτομία σε κάποια συγκεκριμένα κέντρα είναι πολύ σημαντικό γιατί τελειώς θα υπάρχει μεγάλος διασκορπισμός και δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Επίσης, ε, το να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες είναι ζωτική σημασία. Για πολλούς ανθρώπους το να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σε τέτοιο επίπεδο είναι. Είναι πολύ δύσκολο και αν γνωρίζει κάποιον κάποιον που ξέρει πώς γίνεται, έχει καλό, αλλά αλλιώ είναι υπερβολικά πολύπλοκη η διαδικασία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να απλοποιηθεί η διαδικασία και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα στους ανθρώπους που μπορούν να υποφεληθούν από τη χρηματοδότηση. Τρίτον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κινηθούμε προς τη χρηματοδότηση που να βασίζεται στα αποτελέσματα, διότι αλλιώς μεγάλο μέρος της ε, καινοτομίας ε, θα πάει χαμένο, θα έχουμε έρευνα χωρίς καινοτομία, το οποίο δεν ωφελεί και κανέναν. Θα είναι καλό λοιπόν η χρηματοδότηση να βασίζεται στα αποτελέσματα. Όσο μεγαλύτερη απόδοση, τόσο ε, περισσότερη χρηματοδότηση. Και αν δεν έχει κανεί αποτελέσματα, να μην λαμβάνει ε, τη χρηματοδότηση, να λαμβάνει μόνο με πολύ μικρό ποσοστό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τέτοιε προσεγγίσεις, διότι θέλουμε καινοτομία, θέλουμε βιώσιμε θέσει εργασία. Και αυτή είναι η ιδέα που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει άλλο κανεί το λόγο. Κύριε Καντέκ, μήπω θα θέλατε να δευτερολογήσετε, να απαντήσετε στα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Καταρχήν, Χαίρομαι ιδιαίτερως για το ζωηρό ενδιαφέρον που δείχνουν οι συνάδελφοι για τη γνωμοδότησή μου και για τις τροπολογίες που θα καταθέσουν. Μεταφέροντας τα σχόλιά τους σε συγκεκριμένες τροπολογίες που θα εξετάσουμε αργότερα. Διαπιστώνω ότι το θέμα του αποτελέσματος και ο προβληματισμός ως προς το αποτέλεσμα είναι ένα σημείο που μας διχάζει κάπως. Θα το εξετάσουμε και επ' ευκαιρία των τροπολογιών. Οι προτάσεις πάντως των συναδέλφων πολύ πιθανό να συμπεριληφθούν στην γνωμοδότηση, να την εμπλουτίσουν. Θα βρούμε τις κατάλληλες συμβαστικέ προτάσεις όπως προσπαθούμε συνήθως να κάνουμε. Και σας ευχαριστώ. Περιμένω και γραπτός τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Το μόνο που μας μένει να αποφασίσουμε σήμερα είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Προτείνω να την ορίσουμε στις 22 Ιουλίου το μεσημέρι. 22 Ιουλίου το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Γιατί θέλουμε στις 6 Σεπτεμβρίου να υιοθετήσουμε την έκθεση αυτή στη συνεδρίασή μας. Μην ξεχνάτε λοιπόν την προθεσμία για τις τροπολογίες. Ε, παρερχόμαστε στο σημείο 10 γιατί έχει καταφτάσει και ο Λάζλος Σουριάν. Θα του δώσω το λόγο λοιπόν προκειμένου να μας παρουσιάσει εν συντομή την γνωμοδότησή του και τα βασικά στοιχεία της. Έχετε το λόγο κύριε Σούριαν. Ευχαριστώ κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για την πενιχρή κατάσταση του προϋπολογισμού του 2011. Το ΕΚΟΦΗΝ κανονικά θα έπρεπε να έχει οριστικοποιήσει τη, γνώση, τη γνώμη του Συμβουλίου επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι όμως που δεν συνέβη. Το γεγονός ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο οφείλεται στο ότι η συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε στο μεταξύ σε ισχύ. Στην περίπτωση ενός τόσο σημαντικού θέματος, ακόμη και δεν πρόκειται για νομοθετική πράξη με την συνηθισμένη της ε, σημασία. Δίνουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια 8 εβδομάδες προθεσμία για να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Αυτή η περίοδος των 8 εβδομάδων δεν άρχισε με την ε, επίδοση, κοινοποίηση του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα αγγλικά, ξεκινάει να τρέχει η προθεσμία αυτήν των 8 εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση των μεταφράσεων και τη δημοσίευση των μεταφράσεων αυτών. Αυτό μέχρι πρόσφατα. Οπότε δεν αναμένεται καμία επίσημη ε, θέση του Συμβουλίου πριν τις ε, αρχές Αυγούστου. Τώρα πώς θα επηρεάσει αυτό το έργο μας. Φάνηκε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσωπών ότι είχε ήδη διαφανεί μια πλειοψηφία δύο τρίτων στο Συμβούλιο. για την ε, γνώμη αυτή. Οπότε περιμένουμε τη γραπτή μόνο απόφαση που θα υπογράψουν οι Υπουργοί Κοφίν. Τι προβλέπει αυτή η γνώμη του Συμβουλίου τώρα. Είναι το επόμενο σημείο που θα εξετάσουμε. Δυστυχώς ε, δεν ε, προαναγγέλει και πολλά θετικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη ξεκινούν με σημείο αφετηρίας τις ε, χώρες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και αυτό επηρεάζει δυστυχώς αρνητικά τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Υπάρχει μια γενικώ διαπιστωμένη έλλειψη χρημάτων, οπότε οι εθνικές κυβερνήσεις ε, προσπαθούν να περιορίσουν, να συρρυκνώσουν τον προϋπολογισμό όσο μπορούν. Και το δεύτερο σημείο αφορά άμεσα εμάς, γιατί τα κράτη-μέλη ισχυρίζονται ότι το Ταμείο είναι μείον και δεν μπορούν να συμβάλλουν ε, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα οι συνεισφορές για το επόμενο έτος θα είναι χαμηλότερες από αυτές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς στην Επιτροπή μας θα πρέπει να Υποβάλλουμε μια τεκμηριωμένη γνωμοδότηση, γιατί τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμη αποφασίσει για το πώς ε, ερμηνεύουν την κατάσταση. Και μερικές χώρες ε, βρίσκονται σε δινή κατάσταση, όπως η πατρίδα μου η Ουγγαρία, και αυτές οι χώρες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα, υπόσχονται ότι θα βρουν τα κονδύλια για το μερίδιό τους στον προϋπολογισμό, γιατί χρειάζονται τα κοινοτικά κονδύλια για τις επενδύσεις και την ανάπτυξή τους. Αυτή τουλάχιστον είναι η θέση της Ουγγαρίας, αλλά και άλλων χωρών που βρίσκονται σε δίνει κατάσταση. Θα δούμε τι θα πει το Κοινοβούλιο στο τέλος. Εμείς πάντως ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να λάβουμε θέση και να ταχθούμε υπέρ ε, των αρχικών κονδυλίων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως λέγαμε ε, παλιά, να επιβεβαιώσουμε το προσχέδιο. Τώρα έχει αλλάξει η ορολογία, αλλά επί της ουσίας περί αυτού πρόκειται. Θέλουμε αποκατάσταση των αρχικών ποσών της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν χάσουμε τώρα αυτή τη ε, μάχη, Έχουμε προς το παρόν την υπόσχεση του σχεδίου του Συμβουλίου που προβλέπει ότι αν δεν βρεθούν κονδύλια για το Ταμείο Συνοχής, τότε το Συμβούλιο θα τροποποιήσει τον προϋπολογισμό και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τους επαρκείς πόρους για την υλοποίηση των στόχων της συνοχής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και να κρούσουμε και το κόδωνα του κινδύνου στις εθνικές κυβερνήσεις ότι τους τελευταίους μήνες ε, φαίνεται ότι μια τέτοια λύση μάλλον δεν θα είναι εφικτή. Γιατί αν δεν ε, ικανοποιηθούν οι ανάγκες φέτος θα μετακυλιστούν στον επόμενο προπολογισμό. Αυτό έχει συμβεί πέρυσι τουλάχιστον που έχουμε μεταφορά των περσινών αναγκών ε, και ανάγκη ικανοποίηση του από το φετινό προπολογισμό. Η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής μας βρίσκει σύμφωνο σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχω ολοκληρώσει την ανάλυση μου, αλλά έριξα μια ματιά και στην πρόταση του Συμβουλίου και φαίνεται ότι το Συμβούλιο εφάρμοσε πολύ έξυπνη τακτική γιατί περιόρισε τα ποσά πλαίσιο, αλλά αυτές οι μειώσεις σε σχέση με το 2010 δεν είναι τόσο σημαντικές και δίνουν υψηλότερα ποσά. Γιατί αν υπολοιπόταν τον κονδυλίο του 2010, το Συμβούλιο θα διαφωνούσε. Γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργούσε με ένα δωδέκατο του προϋπολογισμού λιγότερο κάθε μήνα. Κάτι που δεν θα έβρισκε σύμφωνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε το Συμβούλιο σκέφτηκε ότι αν με τις προτάσεις για το 2011 αυξήσει ελαφρά τα κονδύλια του 2010, θα μπορούσε να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Πάντως, διαβάζοντας κάποιες μεταφράσεις της γνώμης του Συμβουλίου, μπορείτε να διαμορφώσετε κι εσείς γνώμη και να καταθέσετε και τις τροπολογίες σας. Εγώ σκέφτηκα να καταθέσω με τροπολογία που αν δεν έχει αντίρρηση και η πρόεδρος, θα ήθελα να την υποβάλω την τελευταία στιγμή λαμβάνοντα υπόψη και τη γνώμη των συντονιστών για τα διάφορα πιλωτικά προγράμματα ώστε να υποστηριχθούν αυτά τα πιλωτικά προγράμματα από ολόκληρη την Επιτροπή μας. Εγώ λοιπόν θα καταρτήσω ένα κατάλογο αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων με βάση τη γνώμη και των συντονιστών. Αυτό βέβαια δεν θα επηρεάσει το γεγονός ότι τα πιλωτικά προγράμματα που έχουν υποβληθεί από τους συντονιστές δεν θα είναι νομικώς δεσμευτικά. Πάντως, αν προσθέσουμε όλες τις ανάγκες μας, καταλήγουμε σε πενταπλάσια ποσό από ό,τι υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε και το έγγραφο εργασία ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απαρίθμηση των πρωτοβουλειών που προτείναμε. Και αυτή την πρόταση θα πρέπει να την αντιπαρατάξουμε ως προς την πρόταση βιωσιμότητας, το κατά πόσο θα είναι εφικτή δηλαδή αυτή που θα μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή το καλοκαίρι. Στρέφω την κρυφή ελπίδα ότι μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα υποβληθούν πολλές νέες προτάσεις. Αν κάποιο όμως το επιχειρήσει να καταθέσει και νέε προτάσεις μέχρι το Σεπτέμβριο έντος της προθεσμίας, σας παρακαλώ μην το αμελήσετε και υποβάλλετε σε μένα προσωπικά τις προτάσεις γιατί εγώ θα προλιάνω το έδαφος για τις συνεδρίες των συντονιστών. Κύριε Πρόεδρε, αυτά προς το παρόν, ως προς τη γνωμοδότησή μου. Ο συντονιστής του ΕΛΚ συμφωνεί με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης. Ευχαριστούμε κύριε Σούριαν, ο κύριος Γκοτμάνης. Λυπάμαι που παίρνω συνεχώς το λόγο σήμερα. Ως σκιώδης για την ε, δική μου πολιτική ομάδα για τον προπολογισμό θα ήμουν ε, λίγο πιο αυστηρός σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος ε, Σούριαν. Ποια είναι η πρόταση του Συμβουλίου. Η πρόταση του Συμβουλίου είναι να, να μειωθούν οι πληρωμές για τα ταμεία. Οι δεσμεύσεις θα είναι μηδενικές. Όσον αφορά τις πληρωμές όμως, προβλέπεται μείωση 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, αν δούμε τις περικοπές, κάθε ταμείο και κυρίως τα περιφερειακά ταμεία, 120 μάλλον εκατομμύρια είναι η περικοπή προβλέπεται για το κοινωνικό ταμείο, 129 για τα περιφερειακά ταμεία, 328 για υπόλοιπα ταμεία. Μετά την περικοπή του ενός δισεκατομμυρίου και πάλι οι πόροι θα είναι υψηλότεροι σε σχέση με το 2010. Πολύ σωστά το είπε ο κύριο Σούριαν. Αν δούμε όμως το 2010 και το 2009 θα πρέπει να δούμε ότι το ποσοστό απορρόφησης ήταν πολύ χαμηλό, δύο φορές χαμηλότερο από ό,τι στις προηγούμενες δημοσιονομικές προπτικές και αυτό λόγω της κρίσης. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι οι χώρες προσπαθούν να ανακτήσουν τα όσα χάσανε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και το Συμβούλιο είναι αρκετά διστακτικό. Εμείς θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τη στάση του Συμβουλίου ή όχι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα, γιατί το πρόβλημα είναι ότι οι χώρες θα προσπαθήσουν να αυξήσουν το ποσοστό απορρόφησης. Τώρα είναι η ώρα ουσιαστικά να συσσωρεύσουν τις πληρωμές. Δεν αναφέρομαι στην ανάληψη υποχρεώσεων αυτή τη στιγμή. Η συσσόρευση ανάληψη υποχρεώσεων και η συσσόρευση πληρωμών ουσιαστικά αντιστοιχούν συνολικά σε ένα ποσό που φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Συμβούλιο προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κάνει περικοπές στους πόρους και σύμφωνα με την δική μας Επιτροπή νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί ένα μόνο σημαντικό ερώτημα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε εμείς με το Συμβούλιο να πούμε ότι στάση του υπερβολική. Το Συμβούλιο δεν μας δίνει περαιτέρω πληροφορίες για το τι προτίθεται να κάνει. Η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι ότι προτείνεται απλώς να περικοπούν 1,075 δισεκατομμύρια ευρώ στην κατηγορία 1β. Αυτό είναι το ζήτημα που καλούμεθα να συζητήσουμε εμεί σήμερα και να πούμε τελικά αν συμφωνούμε ή όχι ή αν θα θέλαμε κάποιες μικρότερες περικοπές, Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ. Μία ε, επεξήγηση να δώσω σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γκοντμάνης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε προβλέψεις που στείλανε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση προπολογισμού που κάνει λαμβάνει μικρότερα ποσά και δεδομένα από αυτά τα οποία στέλνουν τα κράτη-μέλη. Αν το Συμβούλιο λοιπόν τώρα προχωρά σε περαιτέρω περικοπές, τότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το προτινόμενο ποσό από το Συμβούλιο είναι πολύ μικρότερο από την προτινόμενη πρόβλεψη των κρατών μελών. Ενδεχομένως να επιστρέφουμε ουσιαστικά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενδεχομένως να ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση. Κύριε Στόιμπερ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κοτμάνης ε, ανέφερε το βασικό πολιτικό θέμα, δηλαδή τι θέση θα πάρουμε σε μια γενική οικονομική και δημοσιονομική κρίση στην ε, οποία τα κράτη-μέλη σημαντικά προβλήματα έχουν ως προς ε, τα έσοδά τους. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει μόνο εξοικονομήσεις στους προϋπολογισμούς ε, των ε, περιφερειών και των ε, κρατών μελών. Θα πρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμβάλλουμε και αυτό είναι σημαντικό επιχείρημα το οποίο δεν μπορώ να απορρίψω. Αυτό όμως που μόλις είπε ο συνάδελφος Κοτμάνης έχει να κάνει με τον βαθμό απορρόφησης τα χρήματα που διατίθενται σε περιφερειακό επίπεδο ε, δαπανώνται. Από ό,τι φαίνεται όχι και υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Έτσι ο βαθμός απορρόφησης διαφέρει ανάλογα με το κράτος μέρος και ανάλογα με τον τομέα. Ε, πιστεύω ότι είναι προβληματικό ότι εμείς ε, ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να απεμπολίσουμε κάποιους πόρους με το επιχείρημα ότι δεν ε, απορροφούνται. Πιστεύω ότι είναι πολιτικά σωστό να επιχειρηματολογήσουμε λέγοντας ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν ε, να περιμένουμε μέχρι να δούμε γιατί δεν έχουν δαπανηθεί τα χρήματα αυτά. Να πούμε δηλαδή ότι περιμένουμε τις σχετικές πληροφορίες. Έχει συζητηθεί και μεταξύ των συντονιστών το να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με τον βαθμό απορρόφησης. Πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε γιατί δεν ταπανήθηκαν οι πόροι αυτοί. Είναι πολύ απλοϊκή η λύση απλά να διαγράψουμε τα κονδύλια αυτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να αναγκάσουμε την Επιτροπή να ε, συνοηθεί με τα κράτη-μέλη για να διαπιστώσει γιατί δεν μπορούν να δαπανηθούν οι πόροι αυτοί. Ο κύριος Προστινάρου. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σούριαν για την έκθεσή του. Στο σημείο 3 αναφέρονται τα πιλωτικά προγράμματα και στα πλαίσια της ε, μελλοντικής πολιτικής για, τα, ε, για τις περιφέρειες. Ε, στηρίζεται η δημιουργία πολιτικού προγράμματος ε, για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της κάποιες περιφέρειας και να αντιμετωπιστεί η απειλή της περιφερειακής ταυτότητας. Μιλάμε για την περιφέρεια του Δούναβη και ο κύριος Σούριαν θεωρεί τα δύο προγράμματα αυτά ε, ότι είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Τρίτον, είμαστε κατά της ιδέας του Συμβουλίου να διατηρηθούν οι υποχρεώσεις αλλά να μειωθεί το επίπεδο των πληρωμών και θα συμφωνούσαμε με την Επιτροπή ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία μείωση στο επίπεδο των πληρωμών και θα πρέπει να αποκατασταθεί το ε, ισχύον ποσό. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι η ιδέα σας είναι η μόνη που μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το 2011 κάποια από τα κράτη θα, ε, θα έχουν σημάδια ανάκαμψης, αλλά χρήματα θα δοθούν κυρίως για μεγάλα έργα που έχουν να κάνουν με την υποδομή και η μείωση της χρηματοδότησης θα ε, έχει σοβαρές επιπτώσεις ως προς την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών μέχρι το 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος ε, δεν υπάρχουν ε, θαυματουργοί τρόποι να ε, πολλαπλασιάσουμε το χρήμα. Θα πρέπει λοιπόν τους πόρους που έχουμε να τους δαπανίσουμε σωστά. Όταν μιλάμε για τις εξοικονομήσεις χωρίς να αναφέρεται το πώς θα γίνουν αυτές, χωρίς εξηγήσει. Δηλαδή αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πιστεύω ότι στην κρίση που, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που βρίσκονται οι περιφέρειες, σημαντικό είναι να μην οπισθοχωρήσουμε. Θα πρέπει επειδή είμαστε σε φάση όπου έχουμε πολλά πολιτικά προγράμματα και στην περιοχή του, Δούναμι, του Δούναβη και τα προγράμματα αυτά χρειάζονται χρήματα, θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα είναι χρήσιμο να ε, συνεχίσουμε να ε, έχουμε τα κονδύλια που είχαμε μέχρι τώρα. Βλέπουμε ότι Μία χώρα όπως η Τουρκία έχει πρόβλημα με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το δικαστήριο επανειλημμένα έχει ε, διαπιστώσει ότι ε, τα χρήματα δεν απανώνται σωστά. Μήπως θα πρέπει τουλάχιστον να μην αυξήσουμε τους πόρους για τα προγράμματα αυτά τα προενταξιακά. τη στιγμή που δεν έχουμε επαρκείς πόρους για τις περιφέρειές μας. Ευχαριστώ, Ιωάχιν Τσέλερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και η γραπτή και η προφορική έκθεση του συναδέλφου Σούριαν ενισχύει ε, ένα αίσθημα δυσαρέσκειας που νιώθω. Τα πράγματα είναι πολύ θολά. Εφόσον το Συμβούλιο δεν εξηγεί την κατάσταση, μπορούμε να συζητάμε, δεν έχουμε όμως καμία ασφάλεια, όσον αφορά τη, καμία βεβαιότητα όσον αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις. Όταν βλέπουμε σταμάτημα των πληρωμών, χωρίς επαρκείς εξηγήσεις, Χθε ανέφεραν αρκετοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, τους ε, Λέει ότι υπάρχουν προβλήματα με, τις, ε, με τη συγχρηματοδότηση. Ε, κάποιοι όμως απάντησαν πολύ ειλικρινά ότι έχουν πρόβλημα όσον αφορά την τεχνογνωσία για τη χρήση των πόρων αυτών. Και γι' αυτό συχνά κολλάει η διαδικασία. Δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε αυτό λοιπόν. Το πώς δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές, τους φορείς που ε, θέλουν να υποφεληθούν από τους πόρους αυτούς. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε σε συνεργασία με την Κομισιόν. Η συζήτησή μας αυτή τη στιγμή ε, κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε τις επιτυχίες που είχαμε μέχρι τώρα στην ε, πολιτική συνοχής. Από την άλλη όμως δεν ξέρουμε εάν ε, στο μέλλον θα συνεχίσουμε να έχουμε τις βάσεις γι' αυτό, δηλαδή την επαρκή χρηματοδότηση, διότι τα κράτη-μέλη που εκπονούν τον προϋπολογισμό τους δεν μας έχουν πει τίποτα σχετικό και επίσης δεν έχουμε και πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο πληρούν τα κράτη-μέλη το σύμφωνο σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της 60 δισεκατομμύρια διαθέτει στα πλαίσια ε, αυτού του προγράμματος που ανέρχεται σε 70 ε, δισεκατομμύρια, από πού θα, 17 ε, δισεκατομμύρια, από πού θα προέρχονται αυτά τα 60 δισεκατομμύρια, δεν το ξέρει κανένας. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το από πού θα προέρχονται τα χρήματα αυτά. Ακούμε κάποιες φημε φήμες για μη δαπανημένους πόρους, για πόρους που δεν έχουν απορροφηθεί. Αλλά όσον αφορά αυτό το σύμφωνο σταθερότητας υπάρχουν και κάποιες ε, υποχρεώσεις εδώ, αλλά θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Αλλιώ μπορεί να έχουμε θεωρητικές συζητήσει σχετικά με το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής ε, και να έχουμε και θεωρητικές επιτυχίες. Εάν όμως δεν γνωρίζουμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη, και μάλιστα από αυτού που... Και μάλιστα αν δεν ξέρουμε αν αυτοί που θέλουν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά ε, μπορούν να τα εφαρμόσουν, ε, τότε η συζήτησή μα δεν θα έχει κανένα νόημα. Θα φύγουμε τώρα διακοπέ, αλλά η πολιτική δεν κάνει διακοπέ. Τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώ στο θέμα αυτό και να το συζητήσουμε το θέμα αυτό με την Επιτροπή. για να μπορέσουμε να ε, έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, από ό,τι βλέπω. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον Λάζλο Σούριαν για να απαντήσει. Thank you very much. Ε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που κάνετε, για τις ε, συμβουλές που μου δώσατε. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις καταργάς προς τον συνάδελφο Γκοντμάνης. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι υπάρχει εδώ πέρα μία αντίφαση. Στη συνέχεια όμως είπατε αυτά τα οποία έλεγα και εγώ, επομένως δεν υπάρχει κάτι με κάποια αντίφαση στις τοποθετήσεις μας. Καμία αντίφαση, πολύ ωραία. Με πολύ μεγάλη σαφήνεια θέστε το ερώτημα το οποίο θέλουμε πραγματικά να θέσουμε. Έχει αποφασίσει πραγματικά η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να υποστηρίξει τα ποσά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των τελικών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ή όχι. Είναι αυτή η στάση λοιπόν της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αν κατάλαβα καλά τους προαλήσαντες, οι περισσότεροι πάνω κάτω πιστεύουν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπερασπίσουμε τα ποσά αυτά. Αυτή είναι άλλωστε και η δικιά μου η θέση. Αναφέρθηκα απλώς στην πιθανότητα να αναγκαστούμε να χάσουμε και κάτι στη τελική ανάλυση, στα πλαίσια διαπραγματεύσεων. Και εσείς πολύ σωστά αναφερθήκατε στις πιθανότητες να χάσουμε ένα ακόμα παραπάνω ποσό. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα με διαφορετική τακτική. Και γι' αυτό το λόγο, το Σεπτέμβριο, ελπίζω ότι τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής μας θα υπερψηφίσουν την προσέγγιση την οποία παρουσίασα εγώ και την οποία παρουσίασε και η Πρόεδρος, ότι δηλαδή η ενδεδειγμένη λύση είναι να υπερασπίσουμε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα είναι σαφές ότι ε, τα τελευταία χρόνια Εξαιτία τη ε, σημαντική ανάληψη υποχρεώσεων ξεκίνησαν πάρα πολλά προγράμματα και τα προγράμματα αυτά θα έρθουν αργά ή γρήγορα και οι πληρωμέ. Η περίοδος λοιπόν 2011-2012 είναι η περίοδος αύξησης των πληρωμών. Επομένως οι που προβλέπει το Συμβούλιο είναι τακτική φύση, θα έλεγα και τίποτα παραπάνω. Πιστεύω όμω ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και σε ένα άλλο μέτωπο. Η, πολιτική συνοχή, η πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι μέρο του προβλήματος, αλλά είναι μέρο τη λύση. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μέσω του οποίου μπορούμε να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση των χωρών, των κρατών μελών. Συνεπώς δεν θα πρέπει να μειώσουμε, αλλά θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους που προβλέπονται για τις πολιτικές αυτές. Η πραγματική βέβαια αύξηση των ποσών δεν είναι δυνατή λόγω των οικονομικών περιορισμών που υπάρχουν. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτά που είπατε κι εσείς, δηλαδή τουλάχιστον τρει προτάσει, του κ. Ντόιτ, μια δική μου πρόταση, μια δική σα πρόταση. Είναι πολύ καλέ και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τις συγκεράσουμε, να τις συνδυάσουμε και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε τελικά σε μία καλή λύση. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, θα καταφέρουμε να επιτελέσουμε ένα καλό έργο, ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε ζωή αν θέλετε στα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι στο στάδιο αυτό η μακροπεριφερειακή πολιτική δεν σημαίνει περισσότερα χρήματα, απέτηση για περισσότερους πόρους. Είναι μια πιο ενδυναμωμένη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για κάτι ακόμα. Όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητα, ή πώς θα πρέπει να ονομάσουμε αυτό το νέο μέσο που έχουμε με τα 60 δισεκατομμύρια, δεν πρόκειται για χρήματα, δεν πρόκειται για κοινοτικού πόρους. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συλλεχθεί από διάφορους πόρους, από διάφορες πηγές και να μπει σε ένα κορβανά. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο κανονικά δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί. Δεν αρκεί όμως να πούμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να γνωρίζουμε σε περίπτωση ανάγκης πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αν ένα κράτος μέλος χρειαστεί να υποστηριχθεί μέσω του νέου αυτού μηχανισμού, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευθυνθεί στις αγορές και θα δανειστεί χρήματα, θα αγοράσει εντό οικών χρήματα από τις αγορές με ένα χαμηλό επιτόκιο. Καθώς η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφώς μεγαλύτερη, η εμπιστοσύνη που έχουν αγορές δηλαδή, από την εμπιστοσύνη που έχουν προς τα κράτη-μέλη. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρει να πετύχει ένα πιο ευνοϊκό δάνειο από ό,τι θα πετύχει ένα κράτος μέλος. Τα χρήματα αυτά συνέχεια θα δοθούν προς τα κράτη-μέλη και όχι τα δικά μας χρήματα από την πολιτική συνοχή. Το σύστημα είναι πολύ περίπλοκο, δεν είμαι σίγουρος ότι και εγώ ίδιος καταλαβαίνω όλες τις πτυχές, πάντως ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ από την πολιτική συνοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί για το νέο αυτό μέσο. Δεν πρόκειται δηλαδή να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που έχουμε εμεί στα δικά μας ταμεία της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ που θίξατε το ζήτημα αυτό, γιατί όντως υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, μια σύγχυση. Ακούσαμε το ποσό αυτό, το οποίο είναι τεράστιο ουσιαστικά 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις αγαπητοί συνάδελφοι και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις, όλες αυτές τις συμβουλές σας, καθώς επίσης και τις τροπολογίες που θα καταθέσετε και κατά αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή μας θα καταφέρει να υποβάλει μια καλή γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστούμε η κυρία Κάλεμπεχ. Ευχαριστώ πολύ. που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω μετά τον εισηγητή. Ε, αυτά που είπατε τονίζουν πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Υπάρχει επιθυμία η Επιτροπή μας να στείλει πριν τις διακοπές ένα σαφές μήνυμα προς τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το μέλλον. Θα υπάρξουν τροπολογίες για πολλά άλλα θέματα, αλλά Διαπιστώνω σήμερα ότι όσον αφορά αυτό το θέμα υπάρχει συμφωνία και πιστεύω ότι θα πρέπει να υποφεληθούμε από τους επόμενους δύο μήνες στις πατρίδες μας ώστε να φροντίσουμε οι περιφέρειες να λάβουν την επαρκή χρηματοδότηση διότι είναι ο, κινητήριος δύναμη της οικονομίας και της απασχόλησης. Η απασχόληση χρειάζεται τους πόρους αυτούς ε, και αν Θέλουμε μια αξιόπιστη πολιτική 2020. Δεν θα πρέπει να πιστοχωρήσουμε και να πούμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και με λιγότερους πόρους. Είναι θολά τα πράγματα, πολλά πράγματα όσον αφορά τα κράτη-μέλη, αλλά σημαντικό θα είναι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας να στείλουμε το μήνυμα αυτό ε, να πούμε δηλαδή ότι ξέρουμε προς τα που θέλουμε να κινηθούν τα πράγματα, ε, εάν θέλουμε να ε, έχουμε κάτι καλό για την οικονομία της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τώρα την προθεσμία για τις τροπολογίες, η οποία είναι πολύ σύντομη, διότι αυτό που δεν είπε ο Λάσλο είναι ότι ως συνήθως το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό για τη διαδικασία του προπολογισμού. Αυτό συνηθίζεται. Είναι λοιπόν πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. 26 Ιουλίου είναι η προθεσμία και να σας θυμίσω ότι θα ψηφίσουμε στις 6 Σεπτεμβρίου. Λάσλο, καταλαβαίνω σωστά ότι θα ψηφίσουμε και τις τροπολογίες σου και τις τροπολογίες για την έκθεσή σου, αλλά θα λάβουμε και απόφαση σχετικά με το πιλωτικό πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό οι συντονιστές να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή, να μιλήσουμε και με τον Λάσλο Σούρια. Είμαστε διατεθμένοι να λάβουμε αποφάσει τον ε, Σεπτέμβριο για τα πιλωτικά προγράμματα και... Μία ακόμα παρατήρηση που έχει να κάνει με τα πιλωτικά προγράμματα. Καταλαβαίνουμε ότι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα επιπλέον άρθρο το οποίο επιβάλλεται στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν ε, ληφθεί αποφάσει. Εμεί προβλέπουμε τη χρηματοδότηση για το ίδιο το πρόγραμμα, αλλά δεν προβλέπουμε την περίπτωση που η Κομισιόν δεν έχει το απαραίτητο δυναμικό και στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα θα αποτύχει. Γι' αυτό λοιπόν όποτε λαμβάνουμε αποφάσεις για νέα προγράμματα θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τρέξει τα προγράμματα αυτά. Είχαμε την περίπτωση της στρατηγικής για τη Βαλτική θάλασσα για την οποία και το Κοινοβούλιο προβλέπει ε, πλέον 20 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ε, κατά τα άλλα θα πήγαιναν στην Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες. Ανταυτού, τα χρήματα δόθηκαν για τις εξωτερικές δράσεις και έτσι ενισχύσαμε στις γειτονικές μας χώρες, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχω λάβει τουλάχιστον. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να φροντίσουμε και την ε, διάρθρωση της χρηματοδότησης που προβλέπεται για τα προγράμματα αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο επί της ουσίας θέμα στην ημερήσια διάταξή μας. Η προθεσμία είναι 26 Ιουλίου το μεσημέρι. Παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε την προθεσμία αυτή. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα είναι Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου. 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, είναι στις 7 το απόγευμα στο Στρασβούργο. 7 με 8.30 στο Στρασβούργο στις 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ κύριε Αντελή. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Μήπως το Σεπτέμβριο θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεταξιολόγηση του προγράμματος Urban. Από ό,τι κατάλαβα, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης συμφώνησε. Μπορούμε να έχουμε την ακρόαση σχετικά με τη μεταξιολόγηση του προγράμματος Urban. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με ακρίβεια. Πάντως σίγουρα μετά το καλοκαίρι θα αφιερώσουμε περισσότερη προσοχή στην αστική διάσταση. Θα οργανώσουμε και δημόσιες ακροάσεις ε, και θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κοινοποιήσει την αξιολόγησή της. Και η Επιτροπή Προϋπολογισμών, αν δεν κάνω λάθος. Ο κ. Τσέλερ το είπε ότι μας λείπουν κάποια στοιχεία. Καλό θα είναι να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς προχωράει η εφαρμογή της πολιτικής και της δημοσιονομικές πτυχές επίσης. Ευχαριστώ. Λύεται τις συνεδρίες, αν δεν υπάρχουν διάφορα. Καταρχήν μην ξεχνάτε τις τροπολογίες. Το επόμενο δεκαήμερο θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και σε αυτές. Κατά του λοιπού, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και ραντεβού το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ και τους Δήμινες και εμείς το ίδιο. Καλό καλοκαίρι.